dice, come, come dice. So, good uh, afternoon everybody. Καλησπέρα σε όλους. Έναρξη της 544ης τακτικής συνεδριάσεως της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Απαρτία λοιπόν. Έχει παραιτηθεί ο Γκαμπριέλε Μπίσοφ. Η κυρία Γκαμπριέλε Μπίσοφ. Εξελέγει ευρωβουλευτής. Παρετήθη. Και φεύγει από την ΣΟΚ και ΡΕΞ, από τα δύο τμήματα. Έχουμε νέο διορισμό στις 6 Ιουνίου. Οι νέοι δεν είναι παρόντε. Ράντε Βράντο Βετ, ομάδα 1, Βουλγαρία αντικαστέ τον Μπόιταν Ντάνεφ, ο οποίος απεβίωσε, θα είναι μέλος της ΕΚΟ και της ΤΕΝ. Παρόντες είναι ο κ. Φερνάντο Βανουέν Μουαρίσιο, Δεκαρβάλιο, ομάδα 2, Πορτογαλία. Μπορείτε να σηκωθείτε να σας δούμε. Καλώς ήρθατε. Αντικαθιστά, ο Μάριο Σάρες θα είναι μέλος της ΝΑΤ και της ΡΕΞ. Και τέλος, εξίσου σημαντικό θέμα, Σοφία Ρέιτζέκερ, ομάδα 2, Αυστρία. Σοφία Ρέιτζέκερ. Εδώ είσαστε. Καλώς ήρθατε. Αντικαθιστά τον Wolfgang Ράιφ και θα είναι μέλος της ΕΚΟ, ΣΟΚ και CCMI. Έχουμε λοιπόν συνεπώς απαρτία, θα εγκρίνουμε το σχέδιο ημερησίας διατάξεως της Ολομέλειας. Δεν βλέπω ενστάσεις ή ερωτήσεις όσον αφορά το σχέδιο της ημερησίας διάταξης. Θεωρείται ως εγκεκριμένη. Θα εγκρίνουμε τώρα τα πρακτικά της τελευταίας Ολομέλειας της 15ης 16 Μαΐου 2018 υπάρχουν αντιρρήσεις δεν βλέπω. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Και πάμε σε ανακοινώσεις του Προέδρου. Ετοίμασα ομιλία μια ώρα, αφού έχουμε χρόνο άλλωστε. Μια ωρίτσα έχω. Δεν αληθεύει αυτό. Ευτυχώς για σας κόλλησα σε μία μία εγκεκριμένη διαδήλωση στο κέντρο της πόλης. Έμπλεξα. Πάνω από μία ώρα έχασα στην κίνηση εκεί. Οπότε, πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρώπη μετά τις ευρωεκλογέ που έχουμε τώρα την Ολομέλεια και πριν από ένα από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, τακτικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια που έχει όμως ιδιαίτερο ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή τη φάση, διότι πρέπει να αποφασίσει στατηγικό θεματολόγιο για την επόμενη πενταετία και υποτίθεται ότι θα λάβει αποφάσεις όπου είναι δυνατόν για τις πολιτικές οροπίες μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων τους επόμενους μήνες και ξεκινώντα από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλοί από εσά θα ήδη σημειώσατε ότι υπήρξαν σχόλια, tweet, blogs και ανταλλαγή απόψεων γενικά και από εκεί ε, φαίνεται ότι όλοι είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Ε, ε μεγάλη συμμετοχή πάνω από 50%, το υψηλότερο ποσοστό την τελευταία 20 ετία, μεγάλη επιτυχία και μπορούμε να είμαστε και λίγο υπερήφανοι λίγο για τη δική μας συνεισφορά ως ε, Επιτροπή. Συμβάλαμε και εμείς αυτό το αποτέλεσμα. Και από ό,τι είδαμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, μοναδικό ρόλο, να δώσει κίνητο στον κόσμο να πάει να ψηφίσει, να πάει στα σοβαρά τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και έχουμε το αποτέλεσμα. Ο θρίαμβος των λαϊκιστικών κινημάτων φοβόμασταν πολύ, τελικά δεν επιβεβαιώθηκε, παρόλο που σε κάποιες χώρες αυξήθηκε η ισχύ τους, αλλά αυτή η βάδα που φοβόμαστε τόσο πολύ, τελικά, βλέποντας τα αποτελέσματα, δεν συνέβη. Θα το δούμε και πώς θα είναι η σύνθεση στις 2 Ιουλίου σε αυτή την αίθουσα του Κοινοβουλίου. Δεν πραγματοποιήθηκε το εκλογικό σώμα θεώρησε ότι έχει πέντε χρόνια για να χτίσουμε την ε, αυριανή Ευρώπη και δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Έχουμε άλλα πέντε χρόνια. Σίγουρα ε, δεν έχουμε εύκολο έργο. Ε, τεράστια επένδυση πρέπει να γίνει. Δέχτηκαν οι πολίτε να επενδύσουν πολλά στην Ευρώπη συμμετέχοντα με τόσο σημαντικό ποσοστό συμμετοχή στι εκλογέ και περιμένουν οι πολίτε συγκεκριμένε αποφάσει και απαντήσει. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, φοβάμαι ότι την επόμενη φορά μετά από άλλα πέντε χρόνια η χιονοστιβάδα εξπρές των λαϊκιστικών, εθνικιστικών ε, κομμάτων θα είναι μια πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο πιστεύω ότι τώρα μπορεί να παίξει μετά από αυτά τα αποτελέσματα πιο επιφανή ρόλο αυτή τη φορά, κυρίως χάρη στην παρουσία των τεσσάρων βασικών φιλοευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων που έχουν ισχυρή παρουσία. Το ΕΛΚ 179 ευρωβουλευτές σοσιαλιστές 153, η πρώην Άλντε και τώρα η Renew Europe άλλαξε όνομα πριν από μερικές ημέρες με 106 και η πράσινη με 75. Οι δύο τελευταίες ομάδες είδαν σημαντική αύξηση όσον αφορά τον αριθμό των εδρών. Συνολικά αυτά τα τέσσερα κόμματα αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα της ε, πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 513 μέλη. Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η τελική συμφωνία στο Κοινοβούλιο στις 2 Ιουλίου, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να σημειώσουμε ότι την τελευταία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, οι ηγέτες των τεσσάρων βασικών πολιτικών δυνάμεων συνυπόγραψαν κοινή δήλωση και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για κοινό πρόγραμμα για το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Πολύ καλό αυτό μήνυμα και περιμένουμε το επόμενο βήμα. Και με την Renew Europe, την συνεδρίαση της ΑΛΤΕ, ε, έχουν εκλεχθεί τώρα οι ηγέτες για την έντολη. Το ΕΛΚ έχει εκλέξει στον κατάλογο της ομάδας, επανεξέλεξε τον Μάνφρεντ Βέμπερ, από την, το ελεύθερο κρατήδιο της Βαβαρίας, Γερμανία, οι σοσιαλιστές χθες την Ράτσα Γκαρσία Πέρες από την Ισπανία εξέλεξαν. Ήταν ήδη ευρωβουλευτής. Σήμερα το πρωί το Renew Europe εξέλεξε τον Τάνσον Τσόλος από την Ρουμανία πρώην α, πρωθυπουργό της Ρουμανίας και επίτροπο και να υπογραμμίσω ότι σε αυτή την περίοδο Πρωθυπουργία της Ρουμανίας ήταν η μόνη κυβέρνηση της Ευρώπης που διόρισε υπουργό για διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τη συμμετοχική δημοκρατία. Είχε διορίσει υπουργό και δημιούργησε τέτοιο υπουργείο. Η Πράσινη ΕΦΑ ήδη αποφάσισαν να διορίσουν, να επανεβώσουν τον Φιλίπ Λαμπέρτ από το Βέλγιο και την Σκά από τη Γερμανία σαν συν συν τον Σμιτ από την από τη Σκοτία σαν πρόεδρο της συνιστώσας ΕΦΑ. Έχουν ηγέτες οι τέσσερις ομάδες, συμμετέχουν πλήρως στις συζητήσεις, στις διαπραγματεύσεις, γεύματα, δείπνα, νυχτερινές συνομιλίες, νυχθημερών συζητούν και ετοιμάζονται για το μεγάλο ραντεβού της πρώτης συνεδριάσεως του Κοινοβουλίου στις 2 Ιουλίου Αύριο, όπως γνωρίζουμε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξεκινήσει τις εργασίες για ένα διήμερο, ούτως ώστε να θετήσει στρατηγικό θεματολόγιο για την επόμενη πενταετία. Επίσης, στο θεματολόγιο, στην ημίσια διάταξη, θα συζητηθεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει να ξαναξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι διαπραγματεύσει το νέο πλαίσιο και το ευρωπαϊκό εξάμεινο, αλλά βασικό σκοπός του Συμβουλίου μετά το άτυπο δείπνο, δύο μέρε μετά τις εκλογές, θα είναι να συναυθεί πολιτική συμφωνία με τις βασική θέση των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, υπάρχουν πολλά προς διαπραγμάτευση και όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμα υπάρχει η δυνατότητα, η πιθανότητα να χρειαστεί ε, άλλη μια έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου στις 30 ε, αυτού του μηνός και 1η Ιουλίου, την ημέρα πριν από την εναρκτήρια συνεδρίαση του νέου Κοινοβουλίου για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που δείχνει τις δυσκολίες επίτευξη συμφωνίας μεταξύ όλων των συνιστοσών ε, μετά τις εκλογές, μεταξύ κυβερνήσεων στο Συμβούλιο ε, και ελπίζουμε ότι τελικά θα συγκεραστούν διάφορες τάσεις και θα καταλήξουν σε σωστή στρατηγική απόφαση λαμβάνοντας υπόψη την ψήφο εμπιστοσύνη που έδωσε το Ευρωπαϊκό Εκλογικό Σώμα και την ανάγκη σαφών επιλογών σύμφωνα με τις, α, την εντολή που έδωσε το εκλογικό σώμα σε αυτή τη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως γνωρίζετε κάποιοι από εσά, Πολλά σχέδια κειμένου κυκλοφορούν σαν αφορά το στρατηγικό πρόγραμμα τις τελευταίες ημέρες, αλλά παρόλο που είναι εμπιστευτικά έγγραφα, δεν υπάρχει όμως κάτι λιγότερο εμπιστευτικό από αυτό που είναι εμπιστευτικό. Είχα τη δυνατότητα να δω ένα κείμενο που συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρία του Συμβουλίου ε, Γενικών Υποθέσεων και αισθάνομαι κάπως απογοητευμένος για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το η ατζέντα για το 2030 δεν έχει επιβεβαιωθεί και είναι το σημαντικότερο ε, θέμα για τα επόμενα χρόνια. Κάποιες αντιπροσωπείες ε, θα συνεχίσουν την προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων. Από ό,τι όμως είδα, από το κείμενο που είδα, η αλλαγή του κλίματος και η πράσινη δίκαιη κοινωνική Ευρώπη τονίζονται στην Ευρώπη, όπως και η προστασία των πολιτών, ε, των θεμελιδών αξιών και των ελευθεριών αυτών και ανάπτυξη ισχυρή οικονομία και η προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων στο παγκόσμιο προσκήνιο. Περισσότερα από αυτά τα θέματα μπορεί να έχουν προτεραιότητα. Έχουμε μεγάλη τεχνογνωσία επί σειρά ετών πάνω σε αυτά και μπορούμε να τα προωθήσουμε και έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε διασυνδέσεις και έχουμε και αντιπροσωπευτικότητα. Όλοι μας περιμένουμε ανυπόμονα τα αποτελέσματα και το τελικό έγγραφο που ελπίζουμε ότι θα εγκρίνουν οι ηγέτες πριν από αύριο βράδυ. Κατά τη διάρκεια της, των της συνεδριάς της τελευταίας εβδομάδας είχαμε συνεδρίαση στη Ρώμη με όλα τα Συμβούλια Κοινωνικά και Οικονομικά της Ευρώπης. Ο Τισιάνο Τρέο ε, μας φιλοξένησε στη Ρώμη και βασικό θέμα των συζητήσεων ήταν το θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης και εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα και υιοθετήσαμε την Παρασκευή στο τέλος της συνεδριάσεως άκρους φιλόδοξα συμπεράσματα και ζητούμε το θεματολόγιο, το πρόγραμμα του 2030 που υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο 2015 από τον ΟΗΕ και που ενεκρίθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Συμβούλιο μάλιστα τον περασμένο Απρίλιο να είναι η αδιαμφισβήτητη βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την επόμενη δεκαετία. Θα συνεχίσουμε να πολεμούμε για αυτές τις προτεραιότητες, δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά άλλο ένα βήμα των εργασιών μας μαζί με τις διάφορες νομοδοτήσεις που έχει εθετήσει η Επιτροπή μας ε, τον τελευταίο χρόνο. Και πριν κλείσω να πω ότι σήμερα το πρωί είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω και να μιλήσω στις Ευρωπαϊκές ημερίδες ανάπτυξης, βασικό θέμα φέτος ήταν η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, ενισχύοντας ε, το θεματολόγιο για τους στόχους της χιλιετίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και να έχουμε νέες συμπράξεις στρατηγικές με την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Και όπως είπα σήμερα το πρωί, σαν Ευρώπη θέλουμε να προτείνουμε αυτά τα θέματα σαν βασικά στοιχεία τη συνεργασία με τι άλλε υπήρου και θα πρέπει να είμαστε συνεπεί σαν Ευρώπη, επιλέγοντα αυτά τα θέματα, θεωρώντα αυτά τα θέματα σαν προτεραιότητά μα. Και βεβαίω, όπω ήδη υπογράμμισα, όλοι είμαστε πεπισμένοι και το πάνελ συμφώνησε ομόφωνα ότι η κοινωνία των πολιτών, ιδιωτικό τομέα, όλοι οι φορεί, όλα τα σχήματα και μορφώματα του διεθνούς προσκυνείου θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των νέων συμπράξεων και συνεργασιών. Διότι το θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης στην παγκόσμια διάσταση αυτής μπορεί μόνο με πολλαπλή συμμετοχή να λειτουργήσει. Όλοι οι φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και όλοι οι εταίροι πρέπει να συμμετέχουν. Σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, που είπα λίγα λογάκια και κλείνοντας Επιτρέψτε μου να εκφράσω θερμό καλωσόρισμα σε πολύ στενό φίλο όλων μας. Και είναι ένα από τους κοσμήτορες, Μπερνάν Μπαταγέ, που υποχρεώθηκε να παραμείνει σπίτι του μετά από μια σοβαρό πρόβλημα. Με τα χαρά σα βλέπουμε ξανά εδώ, εν το μέσο ημών, και προτείνω να χειροκροτήσουμε. τον κύριο Χερνάντες Μπαταγέρ. Λοιπόν, αλλάζω γλώσσα. Πάμε στην έγκριση των γνωμοδοτήσεων με τη διαδικασία άνευ συζητήσεως. Είναι 871 ίδια πρωτοβουλία ευρωπαϊκό πλαίσιο για τι επιχειρήση στην κοινωνική οικονομία άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορία. 158 υπέρ, μία αποχή, 0 εναντίον, ομοφωνία. Εγκρίνεται, συγχαρητήρια, μπράβο. Έγκριση ΝΑΤ 774. Μηχανισμός προστασίας, κοινωνικής προστα... πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παναγιώτης Γκόλφας, συγγητής, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 170 υπέρ. Μία εναντίον, τέσσερι εποχέ εγκρίνεται, συγχαρητήρια. Ψηφίζουμε την γνωμότηση ΕΚΟ 486 σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη, πρώτος απολογισμός, επόμενα βήματα. Πέτρα Ζαράνιτς, Καλιέντο Σόριτς, συγγενής Άρχεται η ψηφοφορία. Can we conclude Πέρας ψηφοφορίας. Γιάτσεκ υπάρχει διαδικαστικό από τον Γιάτσεκ. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Δεν καταχωρήθηκε η προηγούμενη ψήφος μου. Εντάξει, θα το σημειώσουμε, θα σημειώσουμε την ψήφο σας. Δεν σας είδα, συγγνώμη. Πέρας ψηφοφορίας. 179 υπέρ, 8 αποχές, εγκρίνεται η γνωμοδότηση και μία ψήφος υπέρ προστίθεται για την γνωμοδότηση Γκόφα που ενεκρίθη. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους συντάχτες της άλλης γνωμοδότησης. Πριν δώσω την Προεδρία, στην Σαμπέλ Κάνιο και την ευχαριστώ διότι έχω φορτωμένο πρόγραμμα για το απόγευμα. Okay. So, uh, Είχαμε τη δυνατότητα να, να βάλουμε μία από τις πρωινές νομοδοτήσεις απόψε το απόγευμα, να αλλάξουμε σειρά. Έπρεπε να το επαληθεύσουμε. Τώρα μας ήρθαν οι πληροφορίες. Βλέπετε ότι αύριο το πρωί θα έχουμε πάρα πολλά θέματα και έχουμε περιθώρια το απόγευμα, οπότε καλύτερα να βάλουμε κάποια θέματα το απόγευμα σήμερα που έχουμε χρόνο. Η συγγητής έρχεται. Αν συμφωνεί η Ολομέλεια, προτείνω να συζητήσουμε τώρα το 10, 6, 9, Χρήση Λαμπαλών, και να το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα. Το προσθέσουμε το σημείο στην ημερήσια διάταξη και θα αφήσουμε τα υπόλοιπα σημεία όσα εγκρίθησαν Μόνο αυτή την αλλαγή να κάνουμε, αν δεν διαφωνείτε. Δεν να υπάρχει διαφωνία. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Ιζαμπέλ. Και σου δίνω την Προεδρία. Και ευχαριστώ και όλους σας. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη μερίσια διάταξη της ολομέλεια με τις γνωμοδοτήσεις ε, σύμφωνα με τη διαδικασία με συζήτηση. Ξεκινούμε με τη συζήτηση της γνωμοδότησης ε, ΕΚΟ 479 είναι διερευνητική γνωμοδότηση με θέμα την οικονομική σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα εντό των μακροπεριφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στου διακρατικού συνεργατικού σχηματισμού. Συγητή ο Δημήτρη Δημητριάδη. Να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Ο εισηγητή έχει στη διάθεσή του πέντε λεπτά. Κύριε Δημητριάδη, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σα. Συζητούμε εκ νέου στην Ολομέλεια το ζήτημα των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και για μια ακόμη φορά συζητούμε όλα τα προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει όλες αυτές ε, τις ε, δεκαετίες ό,τι αφορά τις Τι είναι όμως ε, το διαφορετικό σε αυτό το έγγραφο που ουσιαστικά πέρασε μια μικρή περιπέτεια, ξεκίνησε ως της ιδέας πρωτοβουλίας και Ξαφνικά, χάρη και στη Ρουμανική Προεδρία, έγινε διερευνητική γνωμοδότηση, διότι η Ρουμανική Προεδρία έθεσε τις μακροπεριφερειακές ε, στρατηγικές και ιδίω ό,τι αφορά την περιοχή του Δούναβη ε, ως υψηλή προτεραιότητα. Υπάρχουν ένα προτεραιότητα μάλιστα της ε, Ρουμανίας και γι' αυτό αποφάσισε το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνική επιτροπή, ε, να ε, κάνει αυτή τη γνωμοδότηση διερευνητική γνωμοδότηση. Για πρώτη φορά λοιπόν εξετάζουμε πάρα πολύ προσεκτικά τα κλάστερ ε, που είναι και μία από τις λύσεις για πολλά προβλήματα τα οποία παρατηρούμε στις ε, στρατικές για τις μακροπεριφέρειες ε, ως ε, ομάδα μελέτης και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Παλμιέρη και με τον Μεντόζα που ήταν πρόεδρος τη ομάδας μελέτης αλλά και όλα τα μέλη βέβαια της ομάδας αυτής γιατί είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε επισκέψεις στη Ρουμανία στο Βουκουρέστι οργανώθηκε μια σημαντική ακρόαση με πολλούς συμμετέχοντες όπως και μια μικρότερη ακρόαση εδώ στις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμη και σε πολλές συναντήσεις συζητήσαμε τις μικροπεριφέρειες και με την Επιτροπή Κρέτσου όλος ιδιαίτερος. Δυστυχώς όμως ε, δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας κυρία Κρέτσου γιατί είχε αντιλημμένες υποχρεώσεις. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα είναι εδώ για να παρουσιάσουμε μαζί την γνωμοδότηση. Δυστυχώς όμως δεν βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Όπως και αν έχει όμως το έγγραφο αυτό, ξετάζει δύο θέματα πολύ προσεκτικά. Το πρώτο είναι τα κλάστερ και βέβαια για μια ακόμη φορά υπογραμμίζουμε τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τη γραφειοκρατία. Με βάση όμως τη δική μου εμπειρία, και επειδή είμαι εδώ και χρόνια μέλος της Επιτροπής αυτής, έχω δει τα προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα είναι η συνδεσιμότητα και η επικοινωνία. Δεν έχουμε ούτε καλή ε, διασύνδεση, καλή συνδεσιμότητα και επειδή γνωρίζω καλύτερα το Ιόνιο και την Αδριατική, μπορώ να σας το πω ότι ισχύει. Ούτε επικοινωνία καλή υπάρχει και το έχω ε, ξαναπεί ενώπιόν σας ε, το θέμα αυτό τη συνδεσιμότητα. Το έχω θέσει και κατά το παρελθόν. Να σας δώσω μια εικόνα. Έχουμε ένα δήμαρχο στο τραπέζι από το Σπλίτα, ένα δήμαρχο από τα Τύρανα και ένα δήμαρχο από το Βελιγράδι. Κάποια μέλη ΜΚΟ από τις χώρες αυτές και κάποιους δημοτικούς συμβούλους ή κάποιους ε, άλλους φορείς και επίσης κάποιους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και προσπαθούν να βρουν ε, κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα να συζητήσουν σημαντικές λύσεις για την περιοχή Αδριατικής Ιωνίου. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση και σχέση μεταξύ φιλοσοφιών και ανατροπιών ε, όλων αυτών. Πώς μπορούμε τι τελείω διαφορετικέ αυτέ προσεγγίσει, φιλοσοφίε να τι προσεγγίσουμε μεταξύ του. Αυτό είναι το πρόβλημα τη μακροπεριφέρειε ε, και ιδίω για το Δούναβι και για την Αδριατική και το Ιόνιο. Καλύτερη εμπειρία ήταν και είναι φυσικά ευαλτική. Βαλτική. Στις Άλπεις επίσης δεν έχουμε τα ίδια προβλήματα που έχουν ε, οι άλλε μακροπεριφέρειες. Και τώρα έχουμε στο χάρτη τη σύνδεση με τη Μαύρη Θάλασσα. Η ομάδα 1 πέρσι είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση για τη Μαύρη Θάλασσα, το Δούναβι και τα συζήτησα αυτά. ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Τώρα θα ολοκληρωθεί εδώ η γενική συζήτηση και το λόγο θα λάβει ο κύριος Μπαράτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη συνάδελφοι και αξιότιμη κυρία Σίτα, ε, θεωρώ πως έχει γίνει εξαιρετική δουλειά σε αυτή τη γνωμοδότηση και όσοι από εσά ε, είχατε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σα για να διαβάσετε αυτή τη γνωμοδότηση, θα διαπιστώσατε νομίζω ότι όλες οι ιδέες ε, που ε, περιλαμβάνονται εδώ βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και καταδεικνύουν δηλαδή ότι χρειαζόμαστε μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Οπότε πραγματικά συγχαίρω τον εισηγητή και τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην κατάρτιση αυτή της νομοδότηση. Ε, σας συγχαίρω λοιπόν ε, για αυτά τα θετικά στοιχεία, αλλά θα ήθελα να ασκήσω κριτική στην Επιτροπή και σε άλλους ε, φόρους ε, διεθνούς πολιτικής σε σχέση με τα όσα κάνουν από τη δική του πλευρά. Και αυτό γιατί δεν αναγνωρίζουν τον ρόλο κλειδί που θα μπορούσαν να παίξουν οι μακροπεριφέρειες. Εάν λάβουμε υπόψη μας τις χώρες οι οποίες συμμετείχαν εδώ και αν λάβουμε υπόψη μας την ε, ιδεολογία η οποία αλλάζει συνέχεια, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής θα μπορούσε να αποτελέσει την απαρχή για ε, τη διασφάλιση μιας σταθερότητας. Θα μπορούσε δηλαδή να ε, ενισχύσει την διασυνοριακή συνεργασία και υπάρχουν μία σειρά από περιφέρειες, μία σειρά από περιοχές στις οποίες η εν λόγω συνεργασία θα μπορούσαν να είναι δυνατή όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τρίτες χώρες. Ε, αυτό δεν αναφέρεται μέσα στη μελέτη αλλά ε, θεωρώ πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιε προσπάθειε οι οποίε γίνονται και για παράδειγμα στην περιοχή τη Μεσογείου, οι οποίε θα πρέπει και αυτέ να λαμβάνονται υπόψη. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δημητριάδη για την επικοδομητική του στάση, γιατί πραγματικά έλαβα υπόψη του όλε τι ε, διαφορετικέ προτάσει. Ο κύριο Μεντόχα Κάστρο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή για την προσπάθεια σύνθεσης ε, και δεν ήταν εύκολο να υπάρχει ένα κείμενο χωρίς τροπολογίες. Ε, νομίζω ότι στην έκθεση αυτή τονίζεται πολύ δικαιολογημένα ε, η σημασία που έχει για τους Ευρωπαίους πολίτες η περιφερειακή πολιτική, η σημασία της ένταξης ε, και της δημιουργίας ε, μακροπεριφερειών και η ανάγκη να πολλαπλασιαστεί το θετικό αποτέλεσμα ε, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της διασυνορικής πολιτικής. Και μετά από 10 χρόνια που έχουμε αυτή τις τέσσερις μακροπεριφέρειες, νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνει ένας απολογισμός ο οποίος και γίνεται με αυτήν την έκθεση, με αυτήν την νομοδότηση, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προκλήσεις για την μακροπεριφερειακή πολιτική, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα, την μετανάστευση, την παιδεία, τα κοινωνικά θέματα κτλ. Επίσης, γίνεται αναφορά σε μια δέσμευση που έχει να κάνει με την αηφορία του περιβάλλοντος και την ψηφιοποίηση Επίσης, αν ληφθεί υπόψη και η στρατηγική 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αυτή η γνωμοδότηση φράζει απαιτήσει ε, και είναι απαιτητική ακριβώς γιατί οι μακροπεριφερειακές ε, στρατηγικές ε, θα πρέπει να εφαρμόσουν στην πράξη την πολιτική δέσμευση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει να οδηγήσουν σε βελτίωση των οργανωτικών κριτηρίων, να δημιουργήσουν μεγαλύτερη διαδικτύωση και να ενισχύσουν το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Πρόκειται λοιπόν για μια ισορροπημένη άρτια γνωμοδότηση ότι αφορά την ανάλυση ε, της πρότασης την οποία διενεργεί και κυρίως ε, λόγω των απαιτήσεων που ε, εκφράζει για ε, το πλαίσιο αυτό. Γιατί πρόκειται για συγκεκριμένα σημεία που μπορούν να δείξουν πάρα πολύ καλά στον πολίτη τι κάνει η Ένωση. Γιατί είναι ακριβώς πιο κοντά σε αυτόν. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, κύριος Πιέτκιβιτς. Σα ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο απλώς ε, για να υποστηρίξω και εγώ εμφαντικά αυτή τη γνωμοδότηση και προκειμένου να κάνω κάποια σχόλια. Έχει καταστηστεί πολύ σωστά αυτή η γνωμοδότηση και λαμβάνει υπόψη ε, τι ε, διεθνεί τάσει που παρατηρούμε. Είχαμε το Παγκόσμιο Φόρουμ χθε και προχθέ ε, στη Γενέβη, όπου συμμετείχαν μέλη διαφορετικών οργανώσεων από ολόκληρο τον κόσμο. Ε, και το ζήτημα της συνεργασίας εντός των περιοχών και αυτή η συνεργατική μηχανισμή, αυτά τα clusters, αναφέρθηκε επανειλημμένα ε, στο Παγκόσμιο Φόρουμ. Και ακόμα και ο keynote ε, speaker, που είναι και ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, τόνισε και εκείνο αυτή την τις πτυχές της παγκοσμιοποίησης που μπορούν να συμβάλλουν σε μια, σε μια πιο συμμετοχική ε, συνεργασία. Άρα λοιπόν αν έγινε ακριβώς αναφορά σε αυτή την υπεραξία των κλάστερς. Και βέβαια εδώ αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους συνεργατικούς ε, μηχανισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παρόλα αυτά η αξία τους ε, αναγνωρίζεται παγκοσμίω. Οπότε πραγματικά σας συγχαίρω για αυτή την γνωμοδότηση. ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να εκφράσω από την υποστήριξή μου, καθώς και της ομάδας μου. Έχουμε διοργανώσει κάποιες εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια, άλλωστε με στόχο την περιφερική και μακροπεριφερική συνεργασία. Το ίδιο κάναμε ε, για τη Μεσόγειο 1 και για το Δούναβι άλλο 1 και επίσης για τη Σαρκία και την Βαλτική 1 τρίτο. Ε, event. Πάντως ε, και οι τέσσερις ε, μακροπεριφέρειες και στρατηγικές, όχι μόνο η Βαλτική, μπορεί να μας δώσει πολλά θετικά. Έχουμε οικονομίες κλίμακας, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να υπάρξει μια μόχλευση των αποτελεσμάτων. Άρα Είμαστε θετικοί απέναντι σε αυτή την προσέγγιση και δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες βέβαια, αλλά θέλουμε να ενταχθούν στον ευρωπαϊκό μηχανισμό υλοποίησης με συμμετοχή κρατών μελών περισσότερων για να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ώστε να έχουμε και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό επιτυχάνεται και με την Ευρωπαϊκή Υποστήριξη. Συγχαρητήρια για την γνωμοδότηση. Εμείς εδώ είμαστε συνεπείς στο ότι υποστηρίζουμε τη μακροπεριφερειακή προσέγγιση. Αυτά ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια. Muchas gracias. Σας ευχαριστώ και σχά, κύριος Χακίν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση. Ήμουνα μέλος της ε, ομάδας μελέτης μου άρεσαν δύο πράγματα όλος ιδιαίτερος, τα οποία θεωρώ πολύ θετικά για τη γνωμοδότηση. Το πρώτο ήταν πολύ ευρεία η προσέγγιση για το θέμα, έγινε δημόσια ακρόαση, πολλοί εμπειρογνώμονες συμμετείχαν σε αυτή την ακρόαση, εισακούστηκε η φωνή τους, συνεργαστήκαμε με αυτούς τους επαΐοντες και ο εισηγητής μας συνεργάστηκε μαζί τους ήμασταν πάρα πολύ ανοιχτοί. Και αυτό δεν είναι τόσο κοινό όταν ετοιμάζεται να συντάσσετε μία γνωμοδότηση. Είναι πολύ καλό που ήμασταν τόσο ανοιχτοί. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, πιστεύω ότι οι μακροπεριφέρειες είναι ένα νέο εργαλείο. Ε, εντάσσουν κράτη-μέλη. Όχι μόνο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσης, αλλά και γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας τρόπος ε, συνεργασίας και προετοιμασίας νέων ε, έργων και προγραμμάτων μαζί. Αναφέρεται στις διάφορες ε, συστάδες συνεργασίας, μορφώματα συνεργασίας, τα clusters, που στόχο έχουν τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Είναι πολύ καλή ιδέα, διότι αυτός ίσως είναι αποτελεσματικότερος τρόπος από ότι πολιτική συνοχής. Εγώ υπερασπίζομαι τις, ε, ένθερμα τις μακροπεριφέρειες, και τις χρησιμοποιώ στα πλαίσια ε, του τομέα προτεραιοτήτων 10 και πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, ο κύριος Πανιέρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Δημητριάδη και τον πρόεδρο της ομάδας μελέτης και όλους που συμμετείχαν στην ομάδα μελέτης διότι σήμερα μας ε, παρουσιάζουν μια έξοχη γνωμοδότηση και με αυτή τη γνωμοδότηση απαντήσαμε πλήρως στα αιτήματα της Ρουμανικής ε, Προεδρίας. Οι μακροπεριφερειακές πολιτικές έχουν δυνατότητες σημαντικότατες σαν μέσο αναπτυξιακό και οικονομικής, κοινωνικής, εδαφικής συνοχής όμως, όπως μας δείχνει και η γνωμοδότηση που σήμερα παρουσιάζεται, τα αποτελέσματα ακόμα είναι πολύ μέτρια. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω το ότι οι μικρομεσές επιχειρήσεις και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις έχουν υποστεί διπλή πίεση και από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και από την παγκοσμιοποίηση σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η κατάρτιση, η συνεχής των εργαζομένων που είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εντός των περιφερειακών αυτών κόμβων, των clusters. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης αυτών των διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης. γιατί αναφέρθηκε στα προβλήματα διασυνδυσιμότητας και επικοινωνίας. Μπορείτε να καταλάβετε πώς αυτά τα προβλήματα έχουν επιπτώσεις, αρνητικές επιπτώσεις και στα clusters των περιφερειακών σχημάτων και στην προσπάθεια που γίνεται να ε, σχηματιστούν ε, υπερπεριφερειακά τέτοια κλάστερ. Ευχαριστώ κύριε Δημητριάδη και ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στην ομάδα μελέτης. Ε, ολοκληρώσαμε τη γενική συζήτηση. Υπήρξαν πολλά σχόλια άκρος θετικά και δίνω το λόγο στον εισηγητή για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τα επενετικά του σχόλια. Ο κύριος Ζεμπάρα τα αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο ξέχασα να αναφέρω. Κατά την Κυπριακή Προεδρία ήμασταν το μοναδικό θεσμικό όργανο το οποίο κατέρτισε μια γνωμοδοτήση ε, σε ό,τι αφορά την μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη Μεσόγειο. Και τότε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας τηλεφώνησε έτσι ώστε να ξεκινήσει ακριβώς μια νέα προσέγγιση σε σχέση με τη Μεσόγειο. Ε, είναι κάτι λοιπόν το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, και συμφωνώ με τον κύριο Παράτ και πραγματικά ελπίζω πως η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει αυτήν την ε, μακροπεριφερειακή στρατηγική στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειο έχει τα δικά τη ιδιαίτερα προβλήματα και τι ιδιαιτερότητέ τη, αλλά ε, πραγματικά νομίζω πω έχει νόημα να ξεκινήσουμε κάτι. Για παράδειγμα έχουμε το μπλε project για τη Δυτική ε, Μεσόγειο και ίσω θα μπορούσαμε λοιπόν να δώσουμε μια <clears throat> συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια και θεωρώ πραγματικά πως οι μακροπεριφερειακές αυτές, αυτά τα κλάστερ μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν πάρα πολύ στην περιφερειακή μας στρατηγική. Δεν υπάρχουν τροπολογίες όσον αφορά τη γνωμοδότηση. Θα περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία η οποία ξεκινάει. Le vote est fermé. Πέρας ψηφοφορίας. 202 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά και δύο αποχές. Εγκρίνεται με πολύ καλό τρόπο, με πολύ ευρία υποστήριξη η γνωμοδότηση. Ζητώ από τον εισηγητή να παραμείνει εδώ, διότι τώρα θα περάσουμε στην γνωμοδότηση ΕΚΟ 489 για το διεθνή ε, ρόλο του ευρώ. Συνεισηγητή είναι και ζητώ από τον εισηγητή τον κύριο Βαν Μπροκντόρφ να έρθει εδώ στο, στο βήμα. Θα δώσω τρία λεπτά στον εισηγητή και τρία λεπτά στον συνεισηγητή για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ε, θα αξιοποιήσω την ευκαιρία να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα τη Μαλτέζη. Αυτή λοιπόν η γνωμοδότηση αναλύει το ρόλο του ευρώ ε, και Πευθύνει μία έκκληση να καταστεί όλο ένα και πιο ισχυρό το ευρώ σε διεθνέ επίπεδο. Παρότι ε, το ευρώ είναι το δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα στις διεθνείς αγορές, δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την ενίσχυσή του και αυτή η ενίσχυση θα πρέπει να λάβει χώρα σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό θα αποβεί ε, προ όφελο των ε, κρατών μελών τη Ευρωζώνης, αλλά και προς όφελος ε, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίοδο, μία περίοδο δηλαδή όπου βλέπουμε να επανεφανίζονται φαινόμενα προστατευτισμού ε, και όπου οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις δείχνουν να έχουν ε, να βρίσκονται σε στασιμότητα, πραγματικά ε, μία τέτοια προσέγγιση, ενίσχυση του ευρώ θα μπορούσε να βοηθήσει σε διεθνές επίπεδο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια έχει και νόημα αυτή η ενίσχυση και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Εφόσον δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ενιαίο και ισχυρό μέτωπο σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν σε σχέση με την κινέζικη, ε, για παράδειγμα, πρωτοβουλία ε, του, ε, ενιαίας, της ενιαίας ζώνης και του ενιαίου προγράμματος, μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα. Είναι λοιπόν να, απαραίτητο να ανταγωνιστούμε το αμερικανικό δολάριο ενισχύοντας τη θέση μας σε τομείς όπως αυτό της ενέργειας και της αεροπορίας. Ταυτόχρονα η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα αυτή της Ευρωζώνης ε, θα πρέπει ε, να ε, επενδύει περισσότερο στις υποδομές, στην εκπαίδευση και γενικότερα σε κοινωνικές επενδύσεις. Θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι υπάρχει ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και να λαμβάνεται κατάλληλα υπόψη η κοινωνική διάσταση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε και κοινωνική σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Κατά τέτοιο επίσης σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ε, την απαραίτητη ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αλλά και της Τραπεζικής Ένωσης, εάν πραγματικά θέλουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της ενίσχυσης του ευρώ. Εάν δεν κάνουμε αυτά τα επόμενα βήματα ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε άλλοι διεθνείς παίκτες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Κίνα θα ε, μας προσπεράσουν. Πράγμα το οποίο θα αποβεί βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφό μου, τον ε, Δημήτρη, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αλεξάνδροφ που συμμετείχε στην κατάσταση αυτής της νομοδότησης. Θα ακολουθήσω και εγώ τον συνάδελφο ο οποίος χρησιμοποίησε τη μητρική του γλώσσα ε, θα ήθελα καταρχήν να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία και τον πρόεδρο της ομάδος και τον κύριο Αλεξανδρόβ για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η γνωμοδότηση αυτή αποτελεί μια πρόκληση, αποτελούσε και αποτελεί μια πρόκληση για την Επιτροπή, διότι ο διεθνής ρόλος του ευρώ αποτελεί ένα, είναι το ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση ε, ήμουνα ιδιαίτερα επηρεασμένος από τα δημοσιεύματα για το ρόλο του ευρώ και μάλιστα κυρίως από τις δηλώσεις του Προέδρου Γιουνκέρ ο οποίος κατ' επανάληψη τόνισε ότι η επόμενη μεγάλη συζήτηση για το ευρωπαϊκό νόμισμα θα είναι αυτή η οποία θα κατευθύνει και το μέλλον του και κάλεσε την, Ευρωπαϊκή, την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει έναν σημαντικότερο ρόλο και να ενισχύσει περισσότερο το ευρώ. Είχαμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων να έχουμε μια για πρώτη φορά κατά την ταπεινή μου άποψη τόσο στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, με συγχωρείτε, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ήρθε στη δική μας διαβούλευση, δεν θυμάμαι πολλές φορές να έχει συμβεί στο παρελθόν, με το Γενικό Διευθυντή Νομισματικών Υποθέσεων και όχι μόνο αυτό, αλλά να κάνει παρατηρήσεις και επί της γνωμοδότησής μας, κάτι που δεν θυμάμαι να έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν ήταν ιδιαίτερα εξαιρετικά χρήσιμη η παρουσία τους αλλά και όλων όσων από τους κοινωνικούς εταίρους συνεισέφεραν στο διάλογο. Το ευρώ θα παίξει κρίσιμο ρόλο τα επόμενα χρόνια εάν κατορθώσει να περάσει στη συνείδηση των διεθνών επενδυτών. Διότι όσα λόγια καλά και αν λέμε στις Βρυξέλλες, όσο και αν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιθυμούν να το στηρίξουν, μόνο οι διεθνείς αγορές θα αποδείξουν ότι το ευρώ είναι ένα διεθνές ισχυρό νόμισμα και υπάρχει μια πολύ απλή εξίσωση. Η απλή εξίσωση λέει ότι το ευρώ θα καταστεί ένα παγκόσμιο νόμισμα όταν θα γίνει το νόμισμα του ενεργειακού τομέα. Εάν στις κατασκευές και στην ενέργεια κατορθώσουμε να υποστηρίξουμε το νόμισμα αυτό και αν οι διεθνείς επενδυτές κατορθώσουν να ζητήσουν να το χρησιμοποιήσουν ως ένα διεθνές εναλλακτικό εργαλείο οικονομικής, νομισματικής πολιτικής, τότε το ευρώ θα έχει καταστεί ένα παγκόσμιο νόμισμα. Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να συζητάμε γι' αυτό, αλλά θα πρέπει συνεχώς να στρέφουμε το βλέμμα μας προς τις αγορές, διότι δεν θα αποφασίσει κανένα ευρωπαϊκό όργανο μόνο του για το ευρώ. Θα αποφασίσουν οι αγορές εάν το ευρώ πραγματικά είναι ή, θα πρέπει να γίνει στο μέλλον το, το αντίστοιχο νόμισμα που είναι το αμερικανικό δολάριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στη συζήτηση επί της γνωμοδοτήσεως. Colin Lustenhauer, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και τον συνεισηγητή. Άκρο ενδιαφέρουσα η γνωμοδότηση. Πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Επιμακρών το συζητούμε και θα παραμείνει επίκαιρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συζητούμε το θέμα του ευρώ να καταστεί σημαντικότερο νόμισμα στο διεθνές προσκήνιο. Σωστά είπαν οι συγητές ότι χρειάζεται ένα σύστημα δημοσιονομικό ε, ε, σωστό και να έχουμε σύγκληση κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Έτσι το ευρώ να έχει κάποια σταθερότητα και να κινείται σε ένα πλαίσιο οικονομικό σταθερό. Αυτό είναι μια ανοιχτή, δεν επιτυγχάνεται και ήταν μία από τις εγενείς αδυναμίες του ευρώ μέχρι τώρα. Πάνω σε αυτό πρέπει να εστιαστούμε. Το είπαν και οι συγγητές αυτό άλλωστε. Στην παράγραφο 4-6 αναφέρονται στη σταθερότητα του ευρώ και αναγνωρίζουν την αυξανόμενη σημασία του ευρώ στη διεθνή σκηνή και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ε, αγορές κεφαλαίων. Οι μικρές εταιρείες χρειάζονται χρηματοδότηση και πολύ συχνά είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση στη διεθνή χρηματαγορά. Είναι, διευκολύνει την κατάσταση του ευρώ διότι μπορεί να μειώσει σημαντικά το κίνδυνο για αυτές τις εταιρείες αντί να χρησιμοποιούν ένα άλλο εθνικό νόμισμα που είναι μικρότερο, πιο αδύναμο. Και ένα άλλο σημείο που θέλω να τονίσω. Πιστεύω ότι όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται το ευρώ σε διεθνέ εμπορικέ συμβάσει. Το είδα ο ίδιο, κυρίω σε εξαγορέ και συγχωνεύσει. Στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο κάποιε από αυτέ οι συναλλαγέ γίνονται ακόμα σε δολάρια, αλλά υπάρχει μια μετακίνηση ε, προς συμβάσεις συγχώνευσης και αγορών εντός της Ευρώπης αλλά και πιο σημαντικό και εκτός Ευρώπης γίνονται αυτές οι ε, διαπραγματεύσεις συναλλαγές σε ευρώ. Αυτό δείχνει ότι αυξάνεται η σημασία του ευρώ χρησιμοποιείται και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από εκεί βλέπουμε τη σημασία που είναι αυξανόμενη. Χρησιμοποιείται και σε διεθνείς συμβάσεις και διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Φιλίπ Buc. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή και τους συνεισηγητές. Ήμουν μέλος ομάδας μελέτης ε, και πρέπει να σας πω ότι οι συζητήσεις ήταν πολύ ανοιχτές και ενδιαφέρουσες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη γραμματεία η οποία οργάνωσε μια εξαιρετικά καλή ακρόαση με όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Αυτό σίγουρα μας διαφώτισε ως προς τη συζήτηση. Για το ευρώ τώρα. Αναμφίβολα είναι και θα παραμείνει, παραμένει μάλλον ένα ισχυρό νόμισμα. Την προηγούμενη πέμπτη, αν δεν απατώμε, η ΕΚΤΑ δημοσιοποίησε την τελευταία ε, πληροφορίες για το ευρώ ως νόμισμα ε, αποθεματικού χάρη και στη Ρωσία που αντικατέστησαν πάρα πολύ μεγάλο ποσό δολαρίων σε ευρώ, 2 Και βέβαια το δολάριο μπορεί να κυριαρχεί ακόμα και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, σε όλο τον κόσμο, αλλά αν θέλουμε εμείς να προδεύσουμε θα πρέπει να κοιτάξουμε προς τα μέσα και όχι προς τα έξω τόσο πολύ. Διότι το νόμισμα είναι η έκφραση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης. Επομένως, θα πρέπει να βάλουμε τον οίκο μας σε τάξη και να προωθήσουμε μια ισχυρή πολιτική ένωση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα τονιστεί η δύναμη του νομίσματος και θα ενισχυθεί και η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα η χρήση του ευρώ στις διεθνές συναλλαγές, ενέργεια, αεροπορία, συγχωνεύσεις, εξαγορές, ευρύτερη ε, αγορά ε, είναι ένα θέμα ε, που μπορούμε να το συζητήσουμε. Και μια τελευταία παρατήρηση, μας το δεύτερο νόμισμα, αλλά έχουμε το ανταγωνιστή μας, ε, την Κίνα, που ανεβαίνει στην τρίτη θέση και μπορεί να μας περάσει. Και πρέπει να παρακολουθούμε και εκεί τις εξελίξεις. Θέλω να ευχαριστώ τον Σύγητη και τους συνεισηγητές. Και τώρα, λέει πρόεδρος, Στέφανο Μάλια. Eh, eh, eh, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον συγητή και τον συνεισηγητή για τη δουλειά που έκαναν σημαντικότατη αυτή η έκθεση σε άκρος επίκαιρο ζήτημα και θα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο θέμα και τα επόμενα χρόνια. Το ευρώ, όπως ξέρουμε, είναι σημαντικότατο νόμισμα παρόλο που υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι δεν θα τα πάει καλά, όμως τα στοιχεία δείχνουν εντελώς το αντίθετο. Ένα από τα θέματα για τα οποία επικρίνεται το ευρώ είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα κοινό νόμισμα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι αυτό αποτελεί αδυναμία, αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επηρεάζει την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν ε, μια δύναμη στις ε, παγκόσμιες αγορές. Γι' αυτό όσο μεγαλύτερη σύγκληση έχουμε και όσα περισσότερα κράτη-μέλη έχουμε που ανήκουν στην Ευρωζώνη, τόσο το ευρώ θα γίνεται και ισχυρότερο, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θα ισχυροποιείται. Όμως, ανησυχώ λίγο και ανησυχώ λίγο για το πολιτικό κλίμα που διαπιστώνουμε ότι υφίσταται σήμερα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, αρκετά ισχυρές δυνάμεις οι οποίες επιμένουν ε, ε, να κινηθούν κατά της ολοκλήρωσης, περαιτέρω ολοκλήρωσης και κινούνται κατά της σύγκλησης. Αυτό με ανησυχεί. Διότι βλέπουμε ότι κάποιες χώρες για κάποιους λόγους αποφασίζουν να μην μπουν στην Ευρωζώνη. Και αυτό είναι επιλογή γίνεται βάση κριτηρίων. Δεν θέλει η χώρα αυτή να συμμορφωθεί με τα κριτήρια τα οποία έχουμε θεσπίσει για να μπει στην Ευρωζώνη. Και ανησυχώ απ' την άλλη για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη σύγκληση έχοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζουμε τώρα ένα δύσκολο πολιτικό κλίμα. Ελπίζουμε ότι αυτή η έκθεση θα τύχει ε, υποστηρίξεως και ελπίζω ότι ο εισηγητής και ο συνεισηγητής θα εξακολουθήσουν να προωθούν την ίδια γνωμοδότηση και μετά την ψηφοφορία. Ελπίζω, ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Προέδρου στο γεγονός ότι ο κ. Σπανιέρη ήθελε να παρέμβει αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει. Ίσως μπορεί να μιλήσει και εκείνο πάνω σε αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Στέφανο. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, ε, κύριο, τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Βόγκφτορφ τον συνεισηγητή και τον πρόεδρο Ζήπκο τη ομάδα εργασία που έκαναν έξοχη δουλειά. Το υπενθύμησε ο κ. Ντεμπούκ. Ήταν, ε, είχαμε ακρόαση υψή του επίπεδου που έλαβε χώρα. Εγώ σας συμβουλεύω να διαβάσετε προσεκτικά αυτή τη γνωμοδότηση, διότι την προσωπεύει ε, ένα ανάγνωσμα που μπορεί να διαλύσει τις αβάσιμες επικρίσεις, τις παράλογες επικρίσεις, τις επιζήμιες επικρίσεις που στερούνται εσδήποτε αληθείας επιστημονικής και που προέρχονται όλο και πιο συχνά επικρίσεις και αφορούν το ρόλο του ευρώ. Μέσω της νομοδότησης η Επιτροπή μας έφερε τη σαφήνεια και εξυπηρετεί ε, την υποστήριξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και του ευρώ αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ λοιπόν τους εισηγητές γι' αυτό. Σα Σας ευχαριστούμε κύριε Παλμιέρη και τώρα έχουμε μια τροπολογία την οποία σχετίζει και συνεχίσεις έχουν ε, αποδεχθεί. Τζον Κόμερ είναι ο συντάκτης αυτής της τροπολογίας. Αν συμφωνείτε όλοι, είμαστε εντάξει, έτσι. Ούτως ή άλλως θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και στον συνεισηγητή για να απαντήσουν. Μάλλον για να ολοκληρωθεί έτσι η συζήτηση. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ κυρία μου. Ε, θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου τη παρεμβάση του. Οι ΜΜΕ σίγουρα θα δραματίζουν ένα βασικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στι ε, χρηματαγορέ και ελπίζουμε ε, να ολοκληρωθεί η Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών, οπότε να μπορέσουν να δανείζονται με χαμηλότερο κόστος, γιατί αυτό θα βοηθήσει σίγουρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν περισσότερο. Φίλιπ Ντεμπούκ μίλησε για ένα πολύ ισχυρό νόμισμα αποθεματικού, αποθεματικό νόμισμα, το ε, ευρώ είναι μια σημαντική εξέλιξη και ο Σπαλμιέρη είπε ότι είναι σημαντικό νόμισμα το ευρώ. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι έτσι να παραμείνει αλλά και να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο και να είναι μεγαλύτερη παρουσία του σε τόμεις όπως η ενέργεια και οι αερομεταφορές. Θέλω να ευχαριστώ και τον Στέφαν για τις παρατηρήσεις του. Και ένα τελευταίο σχόλιο, ναι, πράγματι πρέπει ε, να βάλουμε τα του οίκου μας σε τάξη. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά και στην Ευρωζώνη πολλό μάλλον. Σίγουρα όμως πρέπει να είμαστε και εξωστρεφείς ε, και να υιοθετήσουμε μία ενιαία προσέγγιση, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση και την ε, επιτυχία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Τώρα έπρεπε να είχα πει ε, για την τροπολογία. Είναι μία και μόνη, την έχει δεκτεί ο συγητής και ο συνεισηγητής. Αν συμφωνείτε όλοι, θα και ρίξω την έναρξη της ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Euh, non, c'est pas grave, j'ai le titre Le vote Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται λοιπόν η γνωμοδότηση με 200 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και 3 αποχές. Χαρητήρια. Alors, avis SOC 627, renforcer l'état de... Ενίσχυση του κράτους δικαίου τώρα. Κατέλα, Αντώνιο Μωρίνο Ντίαθ, Καρολίνα Δεσές Μαλέκα. Euh, Είναι η ΣΟΚ 627. Τρία λεπτά για τον κάθε εισηγητή για την περαιτέρω ενδυνάμωση του κράτου δικαίου τη Ένωση. Αποφασίστε εσεί ποιο θα πάρει πρώτο το λόγο. Dziękuję Pani Wiceprzewodnicząca. Szanowni Państwo, będę mówić po polsku. E, chcielibyśmy przedstawić Państwu opinię. Θα τα πω στα πολωνικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μας, η οποία είναι το αποτέλεσμα της εργασίας τριών συνεισηγητών, από τρεις διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Διόλου τυχαίο, καθότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτής της γνωμοδότησης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα ορίσει τις ζωές μας τα επόμενα χρόνια. Μιλώ για το σεβασμό στο κράτος δικαίου. Είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρεται σε πολλές γνωμοδοτήσεις. Μάλιστα συγκροτήθηκε μια ειδική ομάδα για να πραγματευτεί τα ζητήματα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου υπήρξε και μια διαβούλευση της Κομισιόν, απαντήσαμε και εμείς προσπαθώντας να δούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που θα καταστήσουν πιο αποτελεσματικό το σεβασμό του κράτους δικαίου στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάσαμε την ανάλυση και τις υποδείξεις μας ακριβώς για την ενίσχυση, τη βελτίωση των εργαλείων που θα προωθούν ε, το σεβασμό του κράτους δικαίου. Επειδή λοιπόν η Κομισιόν ε, δρομόγησε αυτή την πρωτοβουλία, εμείς θέλουμε να πάρει τακτικό χαρακτήρα, γιατί θεωρούμε ότι ακριβώς οι Ευρωπαίοι, οι ε, συμπολίτες μας που κατοικούν στις πόλεις, στα χωριά, ε, είναι αυτοί που θα πρέπει να αποφασίζουν για το μέλλον. Είναι ενεργετική η προσέγγιση Κομισιόν, proactive, βασίζεται στην πρόθεση του κράτους δικαίου και των αξιών πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στη δική μας γνωμοδότηση τονίζουμε τη σημασία της εκπαίδευσης. Ιδίω τη εκπαίδευσης που ε, απευθύνεται στις νέες γενιές, αλλά και στις δικές μας ηλικίε, στη δική μας γενιά, για να ξέρουμε και εμείς ποιες είναι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένταξης, Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αυτές οι αξίες δεν είναι μόνο οικονομικές, παρότι έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο η οικονομία κατά τη στιγμή της ίδρυσης της Ένωσης, αλλά τώρα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο η μελλοντική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο. Γιατί, διότι είναι οι οργανώσεις που είναι τα πρώτα θύματα καταστάσεων όπου αυταρχικές δυνάμεις, ε, πολιταρχικές δυνάμεις μπορεί να φτάνουν στην εξουσία. Και εκεί ακριβώς, σε αυτό το επίπεδο, επισημένονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, από τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το δίκτυο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Ένα ειδικό λόγιο ένα ετήσιο φόρουμ στο οποίο θα συναντώνται αυτές οι οργανώσεις είναι κάτι πολύ θετικό γιατί εκεί μπορούν να συζητούν τα ζητήματα της επικαιρότητα. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλησπέρα συνάδελφοι. Από δική μου πλευρά θα προσθέσω ορισμένες παρατηρήσεις. Θεωρώ πως το σημείο αφετηρίας τη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα έτσι ώστε να υπερασπιστούμε και να προωθήσουμε το κράτο δικαίου σε όλα τα επίπεδα. Και ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα για να το επιτύχουμε. Άρα λοιπόν, ε, η προστιθέμενη αξία αυτή τη ανακοίνωση είναι ότι ξεκινάει μια ευρία συζήτηση, ένα ευρύ διάλογο για αυτό το θέμα. Ε, ένα από τα κύρια στοιχεία που μας απασχόλησε μας σε αυτή τη γνωμοδότηση ήταν το να διευκρινίσουμε το ρόλο που μπορεί να παίξει η δική μας Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ως ένας από τους φορείς οι οποίοι ακριβώς θα αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για την πρόθεση του κράτους δικαίου. Και επίσης θεωρούμε ότι μπορούμε να ε, αξιοποιήσουμε αυτό το νέο εργαλείο, δηλαδή του ε, μηχανισμού επαγρύπνησης ή εποπτείας του monitoring mechanism. Και τι είναι εκείνο που μας καθιστά διαφορετικούς ως Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε σχέση ακριβώς με αυτό το εργαλείο της παρακολούθησης, της εποπτείας, είναι το γεγονός ότι εκπροσωπούμε την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Όχι δηλαδή μόνο σε εκείνε τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών που εστιάζουν στα ε, ε, ε, ζητήματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά εκπροσωπούμε και του κοινωνικού εταίρου, τι επιχειρήσει και ούτω καθεξή. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έχουμε πραγματικά ένα, μια πολύ ισχυρή βάση και έχουμε μια πολύ ισχυρή φωνή που πρέπει να ακουστεί. Και εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αποκτήσουμε ένα νέο κύρος ως Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και να αναλάβουμε ένα τμήμα από το άχθος των υπολείπων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέει δηλαδή είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο το Συμβούλιο ή μόνο την Επιτροπή. Πρόκειται για κάτι που είναι σημαντικό για όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το γεγονός ότι καθώς εγώ έχω ακριβώς ε, επιχειρηματικό ε, πόβαστρο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το κράτος δικαίου είναι ακριβώς σημαντικό και για τις επιχειρήσεις, για τον επιχειρησιακό τομέα. Και αυτό γιατί. Γιατί αν δεν υπάρχει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, ένα ανεξάρτητος δικαστικό τομέα στα κράτη-μέλη, τότε δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία αγορά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ουσιαστικά το δικαστικό σύστημα αποτελεί το, το, το, το, την προμετωπίδα, θέλετε, εκείνο που προστατεύει ε, το, το, το, την νομοθεσία στα ε, κράτη-μέλη. Και κατά συνέπεια είναι εκείνο που προστατεύει την νομοθεσία στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώ γνωρίζουμε όλοι πως είναι κακή η καιρή για την ποιήση και για τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως και για το κράτος δικαίου. Ποιο θα μα έλεγε ότι θα συζητούσαμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην όαση αυτή που ήταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι πρόσφατα σχετικά. Εγώ προσωπικά ως πρόεδρος ε, για τα, της ομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου είμαι ιδιαίτερος υπερήφανος για την πολύ γρήγορη αντίδραση που είχε η Επιτροπή μας ε, απέναντι στο αίτημα για άνοιξη οριζοντίου διαλόγου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε τη δυνατότητα, την ευελιξία, την ταχύτητα και νομίζω ότι και η έκθεση δείχνει ότι πολύ ξεκάθαρα με διάβγεια ε, και με πολύ ομό περνάμε τα μηνύματα της ΕΟΚΕ και ε, αναφέρουμε τη σημασία της προάσπισης του κράτους δικαίου και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά Λέμε επίσης ότι εμείς οι είμαστε και η φωνή της Οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών και θέλουμε να την προωθήσουμε. Εγώ προσωπικά για αυτά είμαι πολύ περήφανος. Είμαι επίσης περήφανος και από πλευράς τύπου, γιατί στην ομάδα μας αποφασίσαμε να καταθέσουμε μια γνωμοδότηση με τρεις ε, ε και με τρει. Ε, ε, εισηγητές, γιατί θέλαμε να δείξουμε ότι υπάρχει ομόφωνη και συλλογική δέσμευση των τριών ομάδων για την ε, ε, προστασία του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε η φωνή λοιπόν της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και πρέπει να είμαστε και η κριτική φωνή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε πολύ χρόνο. Η κατάσταση σε πολλές χώρες της Ένωσης είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητική πια. Και δεν αρκεί μόνο να λέμε γενικολογίες και να εξηγούμε πώς έχει κατάσταση. Τρεις εισηγητές που είμαστε εδώ θα θέλαμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτον να είχε κάνει ένα παιδαγωγικό διδακτικό έργο, να μας εξηγούσε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πώς είναι δυνατό το 2019 χωρίς μέλη της Ένωσης να παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα. Και δύο, θα μας άρεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είχε κάνει και αυτοκριτική. Τι κάναμε λάθος ή τέλο πάντων τι δεν κάναμε. Και φτάσανε ε, σε αυτή την κατάσταση ε, τα πράγματα. με την πολιτική δράση, με προτάσεις μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή και αυτό κάνουμε με την γνωμοδότηση που σας υποβάλλουμε προς έγκριση σήμερα. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ Χωσέ Αντώνιο και τώρα θα περάσουμε στη γενική συζήτηση. Δύο λεπτά έχετε σας πενθυμίζω. Γεια σε Κράτσικ. Uh, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για μία ακόμη φορά. Να συγχαρώ ειλικρινά τους τρεις εισηγητές κατάφεραν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν ένα έγγραφο που είναι συνεκτικότατο, περιεκτικότατο που τονίζει και τη σημασία του κράτους δικαίου που προφανώς δεν χρειάζεται καν το συζητήσουμε το θέμα εδώ όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό θέμα είναι από διάφορες απόψεις αλλά επίσης εφιστώντας την προσοχή του κοινού στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Μέσω της εντολής που διαθέτει η Επιτροπή μας, είναι σε άριστη θέση, μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο. Πώς να το πω. Να, είναι σαν γέφυρα, χρησιμοποιείται συχνά αυτή η λέξη, αλλά είναι πολύ ενδεδειγμένη η λέξη, να γεφυρώσει το κενό μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων από τη μια πλευρά και με την κοινωνία των πολιτών από την άλλη σε κάποια κράτη-μέλη. Σε κάποια κράτη-μέλη στα οποία η κατάσταση χρήζει προσοχής ή αντίδρασης αναλόγως. Είναι σαφές ότι σαν ένας ευρωπαϊκός θεσμός που υπερασπίζει τη δημοκρατία, την κοινωνία των πολιτών, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ποικιλομορφία, δεν μπορούμε να υποτιμούμε τη σημασία του κράτους δικαίου που εγγυάται την ύπαρξη όλων αυτών των αξιών. Τούτου λεχθέντος πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια ως θεσμικό όργανο. Πρέπει επίσης να ε, κινηθούμε σωστά. Αποδεικνύει αυτή η γνωμοδότηση ότι η δημιουργία του φορέα του οποίου συμπροεδρεύεται ήταν άριστη απόφαση της Επιτροπής μας. Και χαίρομαι και είμαι υπερήφανο που έχουμε σήμερα επιτάπητο σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ και σίγουρα θα την υποστηρίξω αυτή την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κριστιαν Πιετβουλέσκου τώρα. Γεια σας κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να λάβω το λόγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Επιτροπή για την για το κράτος δικαίου που είναι στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Είναι πολύ σημαντική αρχή και αυτή την περίοδο, μάλιστα όπως είπαν και οι συγητές, όπου τίθεται θέμα της, των πολιτικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τίθεται υποπίεση από διάφορες ε, κυβερνήσεις. Χρειάζεται μια προσέγγιση συγκεκριμένη. Σαν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής πρέπει να κινηθούμε, να κινητοποιηθούμε. Γι' αυτό υποστηρίζω το κείμενο με πλήρη εμπιστοσύνη. Αυτή η γνωμοδότηση είναι αποτέλεσμα άριστης προσπάθειας και εργασίας, χωρίς ομάδα εργασίας όπως επεξηγήθη και είμαι πεπισμένος ότι η Επιτροπή θα βρει όλες τις κατάλληλες λύσεις ώστε αυτά τα προβλήματα τελικά να αντιμετωπιστούν με θάρρος και γενναιότητα διότι εδώ χρειάζεται γενναιότητα ε, να κατονομάσουμε τα προβλήματα να δείξουμε ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία ε, ε, είναι απαραίτητα στοιχεία για τις κοινωνίες μας και για τις χώρες μας και ε, να μην, να μην υπάρχει καταπίεση των ελευθεριών αυτών. Υπέχουμε καθήκον να εγγυηθούμε τη σωστή προάσπιση των δικαιωμάτων. Γι' αυτό υποστηρίζω τη γνωμοδότηση και όπως ανακοίνωσαν και οι συγγητές, είμαστε, είμαστε αντίθετοι στις τροπολογίες που υπευλήθησαν στην ομάδα 3 και θα πρέπει να τοποθετηθώ ανοιχτά κατά αυτών των τροπολογιών. Είμαι κατά αυτών των τροπολογιών που ελήφθησαν στην ομάδα 3. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, λες Πιλάσκι. Ο Λέχ Πιλάσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, σε αυτή την επιτροπή μπορούμε να συζητάμε διάφορα πράγματα και να διαφωνούμε, αν θέλετε. Παραδείγματο χάρη, ποια είναι η διάθρωση των φόρων, πώ μπορούμε να πετύχουμε πιο εύκολα τους στόχους τη βιώσιμη ανάπτυξη, πώ θα αυξήσουμε τι αμοιβέ. Όμω ένα θέμα δεν αμφισβητούμε και δεν διαφωνούμε. Ποια είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το θέμα του κράτου δικαίου. Τα θέματα που άπτονται αυτού του δικαιώματο. Αυτή είναι μια άλλη πρωτοβουλία της Επιτροπής μας, αυτή που συζητούμε τώρα, υιοθετήθηκε και το Μάρτιο εγκρίναμε γνωμοδότηση του κυρίου Μόνς η οποία έκανε μια διάγνωση των αιτίων ε, για τα οποία ε, λόγω των αιτίων αυτών δεν γίνονται απόλυτα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάποιες χώρες. Ε, δεν ξεκινάει τώρα αυτή η συζήτηση. Έχει ξεκινήσει από παλιά αυτή η συζήτηση και ελπίζουμε να κρατήσει πολύ διότι συζητάμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτά διακινδυνεύουμε, αυτά κινδυνεύουν δεν θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκαταβατικοί στην προσέγγιση. Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Διαφορετικά δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Εάν κρυβόμαστε, κρύβουμε τα πάντα κάτω από το χαλί, δεν θα γίνει τίποτα σημαντικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση που συζητούμε είναι σημαντικότατη. Και δεύτερον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να απευθύνουν η έκκληση που κάνουν συνταχτέ τη εκθέσεω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντατικοποιήσει τι προσπάθειε, να χρησιμοποιήσει όλα τα κατάλληλα μέσα, τα αναγκαία μέσα, ε, για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Πριν δεν κάναμε τίποτα. Και ξαφνικά ή πετάμε μια χώρα εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω ή κόβουμε του πόρου που διατέτουμε. Φτάνουμε στο άλλο άκρο. Έτσι. Στην τέταρτη παράγραφο τη γνωμοδότηση αναφέρονται διάφορα μέσα, διάφορα εργαλεία πιο μετριοπαθή που θα μπορούσαν να εθετηθούν αμέσω, χωρί να φτάνουμε στα άκρα. Είναι σημαντικό αυτό που είπε και ο προλαλή σα συνάδελφος. Όπως αναφέρει το σημείο 3.7, στη διάγνωση λέμε ότι οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζονται δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Και εγώ είμαι αντίθετο ε, όσον αφορά τις τροπολογίες που ζήτησε η ομάδα 3. Για μία ακόμη φορά δεν είναι απλώς επί χάρτου συνταγές αυτές που διαβάζουμε. Χθες συμμετείχα στη συζήτηση ε, ε, που αφορούσαν έναν επιχειρηματία που συνελήφθη για τρεις μήνες ε, και, και μετά απελευθερώθηκε και μετά ξανασυνελήφθη. Εν τω μεταξύ όμως κανείς δεν κάνει έρευνες για το θέμα του και η εισαγγελία δεν κάνει τίποτα και υπάρχει αυτή η χώρα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και αυτά συζητάμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και αυτό υποστηρίζω την γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ντάσης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή. Πολύ αγαπητή μου πρόεδρος. Ζήτησα το λόγο για να συγχαρώ τους ε, τρεις συζητητές με όλες μου τις δυνάμεις να τους συγχαρώ, διότι βλέποντα την ηλικία μου έχω επίγνωση ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου από τη δημιουργία της πρώτης ευρωπαϊκής κοινότητας αποτελούσε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, σημαντικά χαρακτηριστικά που κατέστησε αυτή την ένωση ελκυστική μέχρι σήμερα. Παρά όλες οι οικονομικές δυσκολίες και άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε το να επικρίνουμε τις, ε, τις εξουσίες σε διάφορες χώρες είναι ένα καθήκον δημοκρατικό θα έλεγα. Να αφήσουμε ελεύθερες τις οργανώσεις τις κοινωνικές των πολιτών που εκπροσωπούν τους μισθωτούς, τους ε, εργοδότες, τους εργαζομένους ή άλλες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός δημοκρατικού καθεστώτος. Λοιπόν, συγχαίρω Πραγματικά συγχαίρω τους τρεις συζητητέ, διότι ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση ζητώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ακόμα ακριβέστερη και θα έλεγα ακόμα πιο αυστηρή όσον αφορά το σεβασμό του κράτους δικαίου και δεν μπορώ να σα κρύψω την έκπληξή μου διαβάζοντας τις τροπολογίες του πολύ συμπαθητικού συναδέλφου Κριστόφ Καμινεύσκη. Το να δεχτούμε την τρίτη τροπολογία του πιστεύω ότι είναι λογική τελική λύση, η τελευταία τροπολογία που έγινε δεχτεί, οι άλλες τροπολογίες είναι ακατανόητε κατά την απόψή μου. Διότι εάν εμείς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν είμαστε σε θέση να τραβήξουμε τα αυτή θα έλεγα εκείνων που ε, κατέχουν την εξουσία περιφερειακή ή εθνική Ποιο θα το κάνει αυτό γιατί αγαπητοί συνάδελφοι γνωρίζετε πολύ καλά η εξουσία είναι πολύ ελκυστική, έχει ζάχαρη και αυτοί που την έχουν στα χέρια τους προσπαθούν να την κρατήσουν πάση θυσία. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η ένωση υπάρχει διότι δεν ανέχτηκε την έλλειψη ελευθερίας, δεν ανέχθηκε την καταπάτηση των δικαιωμάτων των πολιτών, δεν ανέχθηκε το μη σεβασμό του κράτους δικαίου σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω ότι όλος ο κόσμος θα υπερψηφίσει αυτή την γνωμοδότηση ω έχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιώργο. Στέφαν Μπιλτό τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον τελευταίο καιρό αρέσκεται να αναφέρει το κράτος δικαίου και το επικαλείται κατά την άποψή μου λίγο κάπω όμω με συνθήκες ε, μεταβλητή γεωμετρία. Ξέρουμε τι είναι το κράτο δικαίου. Και θα σας δώσω το παράδειγμα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το συνταγματικό μας δικαστήριο αποτελείται από μέλη τα οποία ορίζονται από τις πολιτικές αρχές και μόνο, χωρίς να υπάρχει ε, καμία νομική αρμοδιότητα ή συνταγματική αρμοδιότητα και δυνατότητα προσφυγή. Τα τρία μέλη τα επιλέγει ο πρόεδρο Δημοκρατία, τρία ο πρωθυπουργό, τρία ο πρόεδρο τη Εθνοσυνέλευση και τρία ο πρόεδρο τη Γερουσία. Ε, το όργανο ρύθμισης ε, των μέσων, το αντίστοιχο ΕΣΟΥΡΟΥ ας πούμε, και αυτά ορίζονται από τις πολιτικές αρχές, ο πρόεδρος από τον πρόεδρο της Δημοκρατία και τα άλλα έξι μέλη από τον πρόεδρο της Γερουσίας και τον πρόεδρο τη Εθνοσυνέλευσης. Περιμένω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στραφεί ε, στη ε, δικαιοσύνη για παραβίαση της νομοθεσίας κατά της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ε, γιατί λέμε για την Πολωνία ότι έχει από τη δίαιτα ορίσει το σταματικό δικαστήριο και ότι ο πρόεδρος ορίζεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για την Πολωνία το λέμε αυτό. Για την Πολωνία δηλαδή απαιτούμε να υπάρχουν νομικές ε, δεσμεύσεις ε, και να λαμβάνεται υπόψη, να λαμβάνονται αυτοί οι νομικοί κανόνες υπόψη. Αλλά για το γαλλικό συνταγματικό, μάλλον για το συμβούλιο αυτό, ε, το συνταγματικό της Γαλλίας δεν το απαιτούμε. Άρα ε, υπάρχει μεγάλη ευαισθησία για το κράτος δικαίου όταν δεν είναι ευρωπαϊκές οι κυβερνήσεις, ε, όταν δεν ε, έχουν ε, κάποια διαφωνία και ακολουθούν την ευρωπαϊκή πολιτική δεν τις ε, ενοχλούμε. Άρα κάπως επιλεκτική είναι η προσέγγιση. Εγώ θα ψηφίσω τις τροπολογίες Καμινεύσκη και αν δεν εγκριθούν θα καταψηφίσω και την έκθεση, την γνωμοδότηση. Σε ευχαριστώ Στεφάν. Οι εισηγητές τώρα θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε όλα όσα υπόθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης. Για δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που εξέφρασαν την υποστήριξη τους απέναντι στην νομοδότηση αυτή και ευχαριστώ γενικά όσους πήραν το λόγο. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και βέβαια ε, σε αυτό το πλαίσιο η υποστήριξη δική σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, στη συζήτηση που έγινε δεν ακούσαμε να υπάρχει κάποια ε, ανητική στάση, μια αντίθετη άποψη. Ε, και οι τροπολογίες τις οποίες λάβαμε ευθύ εξ αρχή ήταν τροπολογίες οι οποίες προέρχονται από, τον, από ένα συνάδελφο και τις οποίες έχουμε λάβει υπόψη μας. Θα ήθελα να επαναλάβω κάποια στοιχεία. Η υποστήριξη του κράτους δικαίου δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, να το πούμε έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δηλαδή είναι κάτι το οποίο γίνεται κατά κάποιο τρόπο σιωπηρά μέσα στο χώρο του δικαίου. Και γι' αυτό το λόγο βράχει πρόθεσμα έτσι, σε καθημερινό επίπεδο ίσως να μην είναι τόσο εντυπωσιακό. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν ορισμένες φορές κάποιες τάσεις οι οποίες εμφανίζονται και οι οποίες είναι ανησυχητικές. Και ε, ε, με αυτόν τον τρόπο ελοχεύει ο κίνδυνο κάποια στιγμή να ε, βρεθούμε σε έναν κόσμο ο οποίο δεν θα είναι τόσο ελληνικό και δεν θα είναι τόσο φιλικό απέναντι μα και στα παιδιά μα. Και γι' αυτόν τον λόγο, αυτό που λέω και στου συναδέλφους είναι ότι ακόμα και όταν τελειώνουμε καθημερινά με την εργασία μας και επιστρέφουμε καθημερινά στα σπίτια μας, θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτή την Ένωση θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια δικαιώματα για όλους. Και αυτό επίσης σημαίνει ότι οι αρμόδιοι ε, σε, πολιτικό επίπεδο θα πρέπει και αυτοί να ε, τηρούν και να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες που μας δεσμεύουν όλους. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο αφορά το σύνολο των πολιτών ε, δεν αφορά περισσότερο τη μία ή την άλλη κοινωνική ομάδα, αφορά πραγματικά τους πάντες. Και αυτό βέβαια είναι σημαντικό και για μας εδώ, για τη δική μας Επιτροπή. Και γι' αυτό ακριβώς ε, δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο συνσηγητής. Ευχαριστώ συναδέλφοι και ευχαριστούμε για τα επενετικά σας σχόλια. Ε, το βασικό συμπέρασμα που εγώ άντλω από αυτή τη συζήτηση που έγινε είναι η έμφαση που θα πρέπει να δώσουμε στο μελλοντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Και νομίζω πως πράγματι θα παίξουμε έναν ισχυρότερο ρόλο σε αυτό το τομέα, στο εγγυσμένο. Τώρα, επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως ε, σε ό,τι αφορά την κατανομή του σχετικού άχθου ανάμεσα στα διαφορετικά θεσμικά όργανα της Ένωσης. Διαβάζοντας κανείς την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διαπιστώνω ότι πρόκειται για μια πολύ καλή σύνθεση όλων των εργαλείων που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Και δεν είναι λίγα αυτά τα εργαλεία. Είναι πολλά. Και εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Οπότε ίσως να αναρωτηθεί κανείς ε, ε, τι νόημα έχει να προσθέσουμε ε, ένα νέο εργαλείο, αυτό το εργαλείο παρακολούθησης, αφού υπάρχει ήδη πληθώρα τέτοιων εργαλείων. η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει κάποια πανάκια εδώ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο θα θεσπίσουμε και το οποίο θα επιλύσει ως διαμαγεία όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η συντονισμένη χρήση των πληροφοριών και της γνώσης που έχουμε μπορεί να οδηγήσει ακριβώς στην καλύτερη αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία ακριβώς βρίσκονται στη διάθεση των πάντων. Αυτή είναι νομίζω η γενικότερη εικόνα που θα πρέπει να έχουμε κατά νου για το μέλλον μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την το, την ομάδα εδώ της Γραμματείας για την υποστήριξη που μας ε, παρήχε. Και παρότι γενικότερα δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα για την κατάρτιση νομοδοτήσεων. Σε σχέση με αυτήν είχαμε ακόμα λιγότερο χρόνο και χρειάστηκε καταρχήν να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι απαραίτητο να ζητήσει και τη δική μας άποψη. Και πράγματι στη συνέχεια το αντιλήφθηκε. Και πραγματικά νομίζω πως αυτή η γνωμοδότησή μας θα είναι χρήσιμη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χωσέ Αντώνιο. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της ΕΟΚΕ. Νομίζω ότι ξεκάθαρη είναι η υποστήριξη της Ολομέλειας ΕΟΚΕ στη γνωμοδότηση που σας παρουσιάζουμε και πριν το ξεχάσω θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κλάοντιο Κράτσιο, τον ε, εμπειρογνώμονά μας που για οικογενειακούς λόγους δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ. Θα ήθελα να του διαβιβάσω την ε, αγάπη και την αλληλεγγύη μου. Και θέλω να πω ότι εσείς μπορείτε να είστε ήσυχοι, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Το 2016 ήδη είχαμε εγκρίνει το 2016 μια ε, γνωμοδότηση. Με δική μας πρωτοβουλία προτείναμε τότε τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είχαμε ε, προτείνει ε, το 2016 ήταν το γάντι που ρίξαμε το 2016 και το οποίο το σήκωσε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, θα χρειαστεί να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε το ρόλο μας, το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών ε, για τη συζήτηση ε, για το κράτος δικαίου. Και κάθε μέρα μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε πολλά στις αποστολές που έχουμε στις διάφορες χώρες, στις συνεδριάσεις που έχουμε, στις ε, διάφορες πρωτεύουσες και πόλεις. Και βλέπουμε ότι οι πρώτοι που είναι θύματα παραβία θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακριβώ οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, κοινωνικοί εταίροι. Αυτή είναι τα πρώτα Δεν θα μείνουν μόνοι του όμω. Η ΕΟΚΕ υψώνει τη φωνή της, ε, ορθώνει λόγο και θα στηρίξει τις ανάγκες, ε, τις καταγγελίες ε, αυτών των οργανώσεων. Οι τρεις συζητητές που είμαστε μπροστά σας, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε πάντοτε στο ύψος της δέσμευσης ε, και της ε, υποστήριξης του σεβασμού του κράτους δικαίου και της υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Muy bien, pues... Um, Πολύ ωραία. Εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Για να δούμε λοιπόν σιγά σιγά τις τροπολογίες. Πέντε τον αριθμό τροπολογίες έχουμε. Οι δύο είναι αποδεκτές και οι τρεις όχι. Προς το παρόν θα ξεκινήσουμε την τροπολογία παριθμών 1 για την παράγραφο 3-7 δεν γίνεται δεκτή από τους ηγητές. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καμιέσκη για να μας εξηγήσει την τροπολογία του. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Κρίστοφ Καμινιεύσκη με λένε. Εκπροσωπώ μια οργάνωση μη κυβερνητική. Ετοίμασα τροπολογίες. Ε, είναι ονόματι της ομάδας 3. Δεν είναι δική μου. Ευχαριστώ εκείνους οι οποίοι προφέρουν το όνομά μου παρόλο που δεν είναι Πολωνοί και το προφέρουν σωστά. Γιατί ήθελα να υποβάλω μια τροπολογία σε αυτό το σημείο. Είναι ξεκάθαρο το σημείο όσον αφορά το μήνυμα. Ε, επιστούμε την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα θέματα τα οποία δεν έχει λάβει υπόψη της στην ανάλυση. Αυτό, σε αυτό το τμήμα, στο 3-7-2 δύο αναφέρουμε το θέμα. Στο πρώτο τμήμα, στις πρώτες φράσεις, έχουμε φράσεις παρακινδυνευμένες. Αναφερόμαστε σε, στην προστασία της δημοκρατίας, προστασία του κράτους δικαίου, αλλά όταν θέλουμε να προστατεύονται και στο μέλλον, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν προτείνουμε μέτρα. Σε αυτό το πρώτο τμήμα λοιπόν, εκεί πρότεινα διαγραφή αυτού του τμήματος, διότι ε, περιέχονται δύο επικίνδυνα πράγματα. Το πρώτο, ε, όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα τουλάχιστον, και ζητώ συγγνώμη, Πρέπει να σεβαστείτε ένα λεπτό και έχετε ξεπεράσει τον προβλεπόμενο χρόνο. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε έτσι σχεδόν μονολεκτικά με μια φράση. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι σε αυτό το πρώτο τμήμα μιλάμε για πολιτικές δυνάμεις, για πολιτικά κόμματα ε, που θα έπρεπε να αναλυθούν διότι θέτουν σε κίνδυνο το κράτος δικαίου Υπονομή μου το κράτο δικαίου, αναφέρει εδώ. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ την οποία απευθύνεται αυτή η φράση δεν πρέπει να έχει εξουσίε επαλήθευση και ελέγχου των πολιτικών κομμάτων. Δεύτερο, σε αυτή τη φράση λέμε ότι τα θεσ... οι θεσμοί, οι κυβερνήσει, τα κοινοβούλια κλπ. Διακόπτει η πρόεδρο. Αν πω κάτι τελικό. Λέω ότι οι θεσμοί αυτοί που ανέφερα. Τέλο τέλος πάντων, ήθελα να εξηγήσω. Ευχαριστώ. Ένας από τους εισηγητές έχει το λόγο για ένα λεπτό, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε αρκετό χρόνο, πιστεύω. Και να αφήσουμε τον κύριο Καμινιέτς και να πει δύο κουβέντες παραπάνω. Είναι σημαντικό θέμα. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχουμε το χρόνο αλλά έχουμε και κανόνες. Ένα λεπτό διατίθεται. Εντάξει, λίγο να ξεπεράσουμε το χρόνο, εντάξει, αλλά σχεδόν διπλάσιο χρόνο μίλησε. Μπορούμε να αφήνουμε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά υπάρχουν και κανόνες. Και ο καθένας πρέπει να ρυθμίζει το χρόνο του κατάλληλα. Αυτό πιστεύω εγώ. Είχα ήδη προειδοποιήσει τον ομιλητή ε, σε κάποιο σημείο ότι έπρεπε ήδη να ολοκληρώνει. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξή. Ε, ε, δόθηκε εντύπωση ότι πρόκειται εδώ για μια πρόταση της ομάδας 3. Ναι, συζητήθηκε, 3, συζητήθηκε μεν σήμερα το πρωί, αλλά δεν πρόκειται για κοινή πρόταση από πλευρά τη ομάδα 3. Απλώς το διευκρινίζω. Νομίζω ότι δεν υπήρξε παρεξήγηση. Ο Κρίστοφ Καμινιέσκι το είπε. Τέλο πάντων, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον κύριο Καμινιέτσκι. Εμείς ε, συνεδριάσαμε μαζί με τον κύριο Καμινιέτσκι για μία ώρα και πάνω. Και πρέπει να σας πω ότι οι τρεις συνεισηγητές ε, θέλουμε τη μέγιστη δυνατή συνένεση και επίπεδο συμφωνίας για τόσο σημαντικό ε, θέμα όπως είναι το περιεχόμενο αυτής της γνωμοδότησης. Βέβαια, δεν μπορούμε παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή να είμαστε ατολμοί σε ό,τι αφορά την ανάλυση της κατάστασης που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το 3 παράγραφος 7 ε, ακριβώς αυτό προσπαθεί να κάνει μια ανάλυση του πώς ε, φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση από πολιτικής πλευράς και πώς ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες που νομιμοποιούνται μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών ακριβώς ε, θέτουν υποαμφισβήτηση αυτές τις ίδιες τις δημοκρατικές αξίες. Δεν το λέει ανακοίνωση της Κομισιόν, όμως οι τρεις εισηγητές που είμαστε εδώ θεωρούσαμε ότι πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ότι υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο και αυτό πρέπει να προβληθεί και να επισημανθεί ε, κι ας είναι και μόνο αυτοκριτική. Ε, Ευχαριστώ, Χωσέ Αντώνιο. Να περάσουμε στην ψηφοφορία της τροπολογίας αυτής. Ευχαριστώ, On ferme le vote. Πέρασε ψηφοφορία. 47 υπέρ, 141 κατά, 19 αποχέ. τροπολογία λοιπόν 1 απορρίπτεται. Περνούμε στην τροπολογία περθμών 2. Για το 3, 12. Και είναι μια τροπολογία την οποία αποδέχονται οι τρεις εισηγητές μας. Zgodziliśmy się na to, aby rzeczywiście wykreślić słowa na przestrzegania. Δεχτήκαμε λοιπόν να φέρθουν αυτές οι λέξει. για να προστατεύουμε το κράτος δικαίου κλπ. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που έχουν οι watchdogs, οι οργανώσει λοιπόν, που παρακολουθούν, εποπτεύουν και ενημερώνουν περί παραβάσεων. Όμως έγινε δεκτή η τροπολογία. Σας ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση, λέει Πρόεδρος. Εσείς παρακαλώ, έχετε το λόγο. Είμαστε, είμαι κατά της πρότασης συμβιβασμού γιατί με αυτόν τον τρόπο εξαιρούμε το, τον, τον, τον, ρόλο της, αυτής της οργάνωσης του Watchdog. Και στην δική μου χώρα, στη Ρωμανία, ο ρόλος αυτού του Watchdog είναι ακριβώς η προστασία των ε, δικαιωμάτων, οπότε θεωρώ πως ε, το αρχικό κείμενο είναι ε, το προτιμότερο κατά τη δική μου άποψη, οπότε εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την πρόταση συμβιβασμού. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καμινιές για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Προσπαθούμε εδώ να βρούμε ένα, ε, μια συμβαστική λύση. Ειδικότερα όταν λέμε ότι αυτοί οι οργανισμοί προσπαθούν ακριβώ να υπερασπιστούν τη διατήρηση του κράτου δικαίου. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ποιο είναι ο ρόλο των δικαστηρίων. Ευχαριστώ. Πολύ καλώ. Εκφράστηκαν όλοι, οπότε τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 2 στα 3, 12. Άρχεται ψηφοφορία. We are talking about the compromise. Ζητώ συγγνώμη. Αναφερόμαστε στη συμβαστική τροπολογία γιατί ε, δεν μας απασχολεί πια η τροπολογία η αρχική αφού δεν έγινε δεκτή έτσι, από τους συζητητές. Άρα η ψηφοφορία που κάνουμε τώρα έχει να κάνει όχι με την τροπολογία 2 όπως υποβλήθηκε αλλά με τη συμβιβαστική τροπολογία. Δεν είναι συμβιβαστική, είναι μία τροπολογία, δεν είναι συμβιβασμός. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε τροπολογία έγινε απλά αποδεκτή. Δεν ήταν συμβιβασμό, απλά μια τροπολογία που έγινε αποδεκτή. Τώρα κάποιο απορρίπτει την αποδοχή ουσιαστικά της ε, τροπολογίας και θέλει να τεθεί σε ψηφοφορία. Δηλαδή δεν συμφωνεί με το γεγονός ότι έγινε αποδεκτή αυτή η τροπολογία. Κάποιος είπε ότι είναι κατά της αποδοχής. Το εξήγησε ο Κριστόφ, εξήγησε την τροπολογία του δηλαδή και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο. Ζητώ συγγνώμη που παίρνω το λόγο. Αλλά νομίζω πω αυτό που συνέβη ε, ήταν ότι υπήρξε μια συμβαστική λύση γιατί οι δύο πλευρέ ε, συμφώνησαν σε ό,τι αφορά μια συγκεκριμένη διατύπωση. Αφού λοιπόν έγινε δεκτό με αυτόν τον τρόπο ο συμβασμός, και υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι κατά της συμβαστικής υποτάσεις, τότε ναι, ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε επί της συμβαστικής τροπολογίας και όχι επί της αρχικής τροπολογίας. Νομίζω το καταστατικό μας είναι πολύ ξεκάθαρο σε σχέση με αυτές τις περιπτώσεις. Πρόεδρε, νομίζω πως δεν υπάρχει εδώ ένα ζήτημα επί το οποίο διαφωνούμε. Απλώς κάποιος χρησιμοποίησε την ε, την, την, ε, την, την έκφραση συμβιβασμό. Ε, αλλά ουσιαστικά δεν πρόκειται για συμβιβασμό γιατί μιλάμε για μια ε, τροπολογία, η οποία έγινε μεν δεκτή από του τρει εισηγητέ τη γνωμοδότηση, αλλά δεν έγινε δεκτή από ένα μέλο τη Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή τη Ολομέλεια. Άρα θα ψηφίσουμε επί αυτή τη τροπολογία που έγινε δεκτή από του εισηγητέ και κάποιο την ονόμασε ω συμβιβασμό. Ακριβώ περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι ένα συμβιβασμό, μια τροπολογία είναι. Λοιπόν, αν καταλάβατε όλοι, προσπάσω να το εξηγήσω κι εγώ, αλλά διαβάστε τι λέει. Λέει τροπολογία, τροπολογία που έγινε αποδεκτή. Δεν είναι αποδεκτή όμως πλέον, άρα ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est fermé. Πέρας ψηφοφορίας. Pour 122. 122 υπέρ, 73 κατά, 20 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν τροπολογία 2. On passe maintenant au amendement Προχωρούμε στην τροπολογία παριθμών 3 για το σημείο 5-2. Δεν έχει γίνει αποδεκτή. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Κριστόφ για ένα λεπτό να μας την παρουσιάσει. Κοιτάξτε, λέγα ότι έχω δύο λεπτά. Όσον αφορά αυτό το σημείο, δεν έχω επιφυλάξεις. Η Επιτροπή Οικονομική και Κοινωνική προτείνει την υποστήριξη ενός νέου μέσου, ενός νέου εργαλείου. Δεν έχω πρόβλημα. Να προσθέσουμε όμως ότι κάθε μέσο αυτού του είδους που αναφέρεται σε αξιολόγηση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάθε τέτοιο εργαλείο, μέσο, πρέπει να χρησιμοποιείται συνετά, ούτω ώστε να μην προκαλεί προβλήματα πολιτισμικά ούτε να ε, χειραγωγείται. Υπογραμμίζουμε την πολιτιστική αξία της Ευρώπης. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή. Εάν μου τελειώνει ο χρόνος, πείτε το μου, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, συνεχίζω. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Έχουμε αποδεχθεί τη φράση που τελειώνει μετά τους πολιτικούς στόχους, τελεία. Όμως οι εισηγητές δεν δέχτηκαν την πολιτισμική σύγκρουση, τα πολιτισμικά προβλήματα, τις συγκρούσεις τις πολιτιστικές. Ευχαριστώ πολύ Κριστόφ. Λουκά θα εξηγήσει την άποψη των εισηγητών. Ε, ναι, πράγματι, εμείς οι τρεις εισηγητές απορρίπτουμε αυτήν την τροπολογία. Ε, και αυτό έγινε σε συνέχεια μιας ε, ε, ακράσα και ελεκτρινού συζήτηση που έγινε με τον Κρίστοφ σε σχέση με αυτό το θέμα. Υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ δηλαδή τα οποία δεν μας βρίσκουν σύμφωνο. Καταρχήν το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με προσοχή, όπως λέει η χρήση του μηχανισμού απαιτεί προσοχή. Μα εμείς θέλουμε απλώς να λέμε ότι ο μηχανισμός θα χρησιμοποιείται όπου αυτό χρειάζεται, όχι με προσοχή. Και μετά το δεύτερο στοιχείο με το οποίο δεν συμφωνούμε είναι αυτή η, ε, η διαφορετική ερμηνεία αν θέλετε των πολιτικών ε, της πολιτικής κουλτούρας αν θέλετε ε, και το ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε, σε πολιτισμικές σύγκρουσεις ε, αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνος ως δήλωση γιατί θεωρούμε πως έρχεται σε αντίθεση με το βασικό μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία. 3. Παράγραφος 5.2. Άρχεται η ψηφοφορία. Le τη est euh, υπέρ 42, κατά 153, αποχές 23, απορρίπτεται η τροπολογία. Πάμε τώρα στην τροπολογία 4 που είναι σχετική με την παράγραφο 1 1-6, που επίσης ε, απορρίπτεται. Ο λόγος ξανά στον Κριστόφ για να μας εξηγήσει την τροπολογία του. Όχι, δεν θα περάσουμε ξανά. Έχω το λόγο ή όχι. Εάν είναι το ίδιο, δεν πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Ήδη απερίφθη η τροπολογία. Ευχαριστώ, Γιώργο. Τροπολογία 5, 1, 11. Σημείο 1, 11. Τροπολογία που έγινε δεκτή. Κυρία Πρόεδρε, με κατά τροπολογίας, διότι η δημοκρατία είναι φιλελεύθερη. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που λένε ότι η δημοκρατία, η φιλελεύθερη είναι πολύ σημαντική, πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Η δημοκρατία είναι φιλελεύθερη. Είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίζουμε αυτό. Και γι' αυτό είμαι κατά. Κριστόφ, ένα λεπτό. Συμφωνώ με τη θέση ότι η δημοκρατία είναι φιλελεύθερη. Αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ φιλελεύθερης δημοκρατίας και του γεγονότος ότι η δημοκρατία είναι φιλελεύθερη. Η δημοκρατία θέλει να είναι φιλελεύθερη, άλλο αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία επιτρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Πρόκειται περί θέματος σημαντικότατου σε αυτό το σημείο είναι θέμα διαφύλαξης της δημοκρατίας να διατηρηθεί το πνεύμα και η καρδιά της δημοκρατίας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Είτε έχουμε δημοκρατία, οπότε την υπερασπιζόμαστε και αν πρέπει να την καθορίσουμε, να την καθορίσουμε την δημοκρατία, τότε αυτό γεννά το κίνδυνο κάποιας διαφοροποίησης και παρεξηγήσεων και παρανοήσεων. Ευχαριστώ. Χωσέ Αντώνιο, ως εισηγητής, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι είχαμε τις αμφιβολίες μας οι τρεις εισηγητές ε, να αποδεχθούμε ή όχι αυτήν την τροπολογία, όμως τελικά ακούγοντας ε, και τις εξηγήσεις ε, είπαμε ότι ίσως καλό είναι να μην δώσουμε ένα χαρακτηρισμό ε, στη δημοκρατία και να μην πούμε σε μία μάχη ε, γλωσσική και ενοιολογική Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ε, στιγματίζουν ε, τη δημοκρατία ανάλογα με τις φιλοδοξίες τους, τον προσανατολισμό τους ε, και τις βάζουν επίθετα και ποιοτικού χαρακτηρισμούς. Μία είναι η δημοκρατία. Οι αξίες, οι αρχές τις περιλαμβάνονται στο άρθρο 2. Και αυτή η έννοια της δημοκρατίας είναι κάτι κοινό για όλους τους πολίτες της Ένωσης και πρέπει να το έχουμε στην καρδιά μας. χωρίς προσδιορισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε λοιπόν την υπαρθμόν 5 τροπολογία για την παράγραφο 1.11. Άρχεται η ψηφοφορία. Se cierra Πέρας ψηφοφορίας. 119 υπέρ, 73 κατά, 21 αποχές, η τροπολογία 5 εγκρίνεται. Και τώρα μπορούμε πλέον να, να ψηφίσουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Eh, Πέρας ψηφοφορία. 190 υπέρ, 11 κατά, 12 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση. ΣΟΚ 627 συγχαρητήρια στους εισηγητές. Και προχωρούμε στην τελευταία για σήμερα γνωμοδότηση. 10692. Ρέιμον Χένξ, ο εισηγητής. Στάνισλαβ Μπάλον, συνεισηγητής. Παρακαλώ, ελάτε στο βήμα. Να ακούσουμε την παρουσίαση της ε, γνωμοδότησης από τους ηγητές. Τρία λεπτά ο καθένας. Παρακαλώ, ξεκινήστε. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή μας έκανε πολλές προσπάθειες για να υπάρχει μια ευρωπαϊκή βάση των κοινωνικών δικαιωμάτων και γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτή τη βάση, αυτό πλαίσιο, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ούτως ώστε 20 αρχές οι οποίες αναφέρονται και διακηρύσσονται να εφαρμόζονται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υλοποιούνται στην πραγματικότητα κάτι που δεν ισχύει για την ώρα. Με αυτό το πνεύμα κινηθήκαμε. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή, έχει 21 αρχές αυτή η γνωμοδότηση. Δικαίωμα πρόσβασης στις βασικές ποιοτικέ υπηρεσίες και αυτές οι θεμελιώδεις υπηρεσίες είναι μια νέα έννοια, βασικές υπηρεσίες που δεν υπάρχει στις συνθήκες. Αν διαβάσουμε τον κατάλογο το μη εξαντλητικό παραδειγμάτων αυτών των υπηρεσιών που παρατίθενται στην 21η αρχή, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται περί υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, είδωρ, ε, υγεία, ε, ενέργεια, αποχέτευση και τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτή αυτή η 21η αρχή επιβεβαιώνει τα ήδη υπάρχοντα, διότι αυτέ οι υπηρεσίε ήδη καλύπτονται από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, από το άρθρο 14 τη συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και από το πρωτόκολλο 26 όσον αφορά τι υπηρεσίε κοινού συμφέροντο. Όμω, αυτό το πρωτόκολλο όσον αφορά τι κοινοφελεί υπηρεσίε προχωρά πιο μακριά από τη 20η αρχή διότι καλεί τα κράτη-μέλη να φροντίσουν να υπάρχει υψηλό ποιοτικό επίπεδο και να υπάρχει ασφάλεια και να μπορεί να υπάρχει προσβασιμότητα, να υπάρχει ισότητα και να υπάρχει καθολική δυνατότητα παροχής, όμως σε κάποια κράτη-μέλη κάποιες υπηρεσίες κοινοφελής δεν ανταποκρίνονται ή ατελώς ανταποκρίνονται σε αυτά τα κριτήρια τα οποία βρίσκονται στο πρωτόκολλο. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να εγκρίνουμε το ότι το πρωτόκολλο επιβεβαιώνει ότι οι βασικές αυτές οι ουσιώδεις υπηρεσίες θα πρέπει να στη διάθεση του καθενός όμως αυτό δεν αρκεί μέσω διακηρύξεως, θα πρέπει να ακολουθηθεί μέσω διευκρινήσεως της ενίας αυτών των ουσιοδών βασικών υπηρεσιών, κάτι που δεν υπάρχει στις συνθήκες και με συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση των υφισταμένων ελλείψεων και να υπάρχει εγγύηση εύρυθμης παροχής των υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Λοιπόν, να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα όπου το πρωτόκολλο 26 προβλέπει ότι θα υπάρξει υπηρεσία ποιοτική αν πάρουμε τις τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Υπάρχει μια οδηγία που αναφέρει ότι κάθε τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Όμως ξέρετε όσον αφορά την κινητικότητα, τα κινητά τηλέφωνα υπάρχουν περιοχές που δεν συνδέονται καθόλου και αυτές που είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο πολύ συχνά η σύνδεση αυτή είναι πολύ μέτρια με το διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα αυτού που αναφέρουμε σε αυτή την έκθεση. Κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς να καλυφθούν αυτά τα κενά και ελλείψεις αλλά εφόσον ξεπέρασα το χρόνο μου θα δώσω το λόγο στον συνεισηγητή για να συνεχίσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω λίγα σχόλια και εγώ γιατί η συνάδελφη ουσιαστικά τα είπε όλα, τουλάχιστον εκείνα που είναι σημαντικά. Ε, να προσθέσω κάτι. Ε, η αρχή 20 του πυλώνα των διωμάτων της Ένωσης ε, αναφέρεται ακριβώς σε αυτές τις ε, υπηρεσίες ε, γενικού συμφέροντος, αλλά αναφέρει επίσης ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη. Και νομίζω πως αυτή η φράση είναι πολύ σημαντική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να είναι υπεύθυνα για την παροχή αυτών των βασικών υπηρεσιών ή ε, αυτών των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος στους πολίτες τους, αλλά, αλλά το γεγονός ότι έχει περιληφθεί πλέον στον, ε, στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων αυτή η φράση συνεπάγεται ότι η παροχή λοιπόν ε, αυτών των υπηρεσιών σε εκείνους που έχουν ανάγκη θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο πλέον και παίζει σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα ακόμα σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Και το γεγονός ότι αυτή η πρόσβαση αποτελεί ένα αναπόσταστο τμήμα της κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απαραίτητο για την Ένωση αφού απαγορεύει οποιοδήποτε είδους δυσμενούς διάκριση ή ή αποκλεισμού, αφού η βασική αρχή είναι ακριβώς αυτή η βασικη αρχη ειναι ακριβω πρόσβαση σε αυτέ τι υπηρεσίε, σε προσιτές ε, τιμέ και με την κατάλληλη ποιότητα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ε, σημαντικό που το τονίζουμε στην δική μα γνωμοδότηση και νομίζω πω ε, περνάμε ένα ισχυρό μήνυμα και προ τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και προ του πολίτε μα και ευχαριστώ πολύ και τον συγητή για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Δεν ζητάει κάποιος το λόγο. Όλα υπήρξαν σαφέστατα και πιστεύω ότι η υποστήριξη θα είναι αρκετά ευρεία. Ξεκινάει ψηφοφορία ε, για το τέν 692. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 128 ε, υπέρ, 6 ε, αποχές και 3 ψήφοι κατά. Υιοθετείτε λοιπόν η γνωμοδότηση και συγχαρητήρια. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις σημερινές μας εργασίες. Θα ξαναρχίσουμε αύριο στις 9.30 το πρωί. Να επενθυμίσω ότι εξαχθεί συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνο για την Ενεργειακή Ένωση. Καλό σας βράδυ. Τα ξαναλέμε το πρωί 9.30. Ευχαριστούμε τις ευχαριστούμε και εμείς που μας ακούσατε. Καλό βράδυ.